Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσουμε την ακρόασή μας και θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους και όσες είναι εδώ. Λυπάμαι, ορισμένες πολιτικές ομάδες το ζητούν ιδιαίτερα για παρόμοιες ε, οργανώσεις, παρόμοια θέματα, αλλά μετά τι γίνεται όσον αφορά την παρουσία τους, τη συμμετοχή τους στην εργασία μας, ε, δημιουργούνται ερωτηματικά. Ίσως ε, στο γραφείο τους ε, είναι αρκετά μέλη και κοιτάνε στην οθόνη της τηλεόρασής τους, είναι συνδεδεμένοι με την αίθουσά μας εδώ και μας βλέπουν από την, ε, από την οθόνη. Έχουμε λοιπόν να συζητήσουμε για τις ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειες σε επιχειρήσεις διαχείρισης διεθνούς κρίσης και όσα γίνονται σχετικά με στα θέματα ασφάλειας και κίνης άμυνας και είναι και επίκαιρο το θέμα, ίσως όχι άμεσα επίκαιρο αλλά τουλάχιστον τελευταίους μήνες και χρόνια. Τι παρατηρήσαμε ότι η χρήση παρομοίων εταιριών στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν αντιμετώπισε και αντιδράσεις βέβαια και αυτό επειδή δεν υπήρχε ένα νομικό σαφές πλαίσιο σε διεθνές επίπεδο για να δούμε τι καθεστώς θα είχαν αυτές οι εταιρείε στα πλαίσια της άσκησης των δραστηριοτήτων τους και στην Ευρωπαϊκή Ένωση η χρήση παρομοίων ε, ε, μέσων ήταν κάπως περιορισμένοι, αλλά επειδή υπήρχαν αρισμένες ε, δυσκολίες στον προϋπολογισμό και επειδή δεν υπήρχε πολιτικό προσωπικό το είπαμε και σήμερα το πρωί άλλωστε για τη Βοσνία και το Κωσυφοπέδιο σε επιχειρήσεις εκεί ίσως το μέλλον και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, την ελκύσει μια παρόμοια δυνατότητα για αυτό το ιδιωτικό προσωπικό της ιδιωτικές εταιρείε. Ε, τώρα τελευταία να αναφέρουμε, θα τα πούμε ξανά σε λίγο, είναι ένας κώδικας διεθνούς συμπεριφοράς που προσυπέγραψαν αρκετές ε, ιδιωτικές εταιρείε ασφάλειας παγκόσμιο, σε παγκόσμιο επίπεδο και που συνεχίζουν να προσυπογράφουν και άλλες και θα προσπαθήσουμε να λύσουμε όσο γίνεται καλύτερα και περισσότερο αυτές τις δραστηριότητες. Έχουμε τρεις ομάδες ομιλητών σήμερα ε, σε τρία μέρη. Πρώτο μέρος ε, με τρεις εμπειρογνώμονες θα σας παρουσιάσω και που θα μας πούν πως έχει κατάσταση πάνω σε αυτό και ακαδημαϊκά, ας το πούμε έτσι, ε, από νομικής πλευράς να δούμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε και επίσης μια δεύτερη ομάδα που θα ακούσουμε έτσι και όσους είναι επιτόπου δηλαδή ορισμένες εταιρείε, όπως τον κύριο Μπέρπαρκ ο οποίος θα είναι εδώ για από την Βρεταϊκή Ένωση των Ιδιωτικών Εταιρείων Ασφαλείας και τον Μάικλ Κλάρκ ε, του G4S των ε, παρομοίων ε, θεμάτων και ένα τρίτο πάνελ με εκπροσώπους υπεύθυνους από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε εξωτερικές ενέργειες, τον κύριο Κλόπενχάουβερ, ε, του CPCC διευθυντή, τον γνωρίζουμε πολύ καλά, και τον Πάτρικ Σάλτ που είναι στη διοίκηση και στα οικονομικά θέματα και που υπογράφουν τα συμβόλαια, τις συμφωνίες σχετικά με τη χρήση παρομοίων ε, εταιριών, χρησιμοποίηση αυτών σε επιχειρήσεις διαχείρισης διεθνούς κρίσης. Ξεκινάμε με την κυρία Αν Μαρή Μπουζατού, συντονίστρια του προγράμματος ε, για την ιδιωτικοποίηση της ασφάλειας, το ε, ε, δημοκρατικό έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων ε, DCAF στην Γενέβη είναι η έδρα, έχει παίξει ενεργό ρόλο και είναι εμπειρογνώμων αναγνωρισμένη στον τομέα αυτό. Επίσης ο καθηγητής κ. Ροντζίτη, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στη Ρώμη και επιστημονικός συνεργάτης και σύμβουλος στο Κέντρο Διεθνών Υποθέσεων και ο κ. Μπράνοβιτς, συνεργάτης στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου γνωστός και εκείνος. Η κυρία Μπουτζάτου έχει το λόγο ξεκινώντας. Στη συνέχεια θα έχουμε και τις υπόλοιπες παρεμβάσεις και μια συζήτηση με τα παριστάμενα εδώ μέλη. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που με προσκαλέσετε να παρουσιάσω στην Υποεπιτροπή του Κοινοβουλίου για θέματα ασφάλειας και άμυνας τις βασικές προκλήσεις σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση των, τους κανονισμούς στον τομέα της παροχής υπηρεσιών στον τομέα ασφαλείας. Θα σας μιλήσω για μια διαδικασία για το πώς ε, μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη λογοδοσία και εποπτεία ε, του ιδιωτικού τομέα παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στο πλαίσιο του Εθνούς Κώδικα Διοντολογίας. Έπειτα θα αναφέρω κάποιες συστάσεις ε, για την Υποεπιτροπή και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε. Σε ό,τι αφορά λοιπόν ε, τις προκλήσεις που τίθενται για τις ιδιωτικές ε, εταιρείες παροχής ασφάλειας, ε, θα ήθελα να αναφέρω καταρχάς, για να τα εντάξω και στο πλαίσιο της συζήτησης, κάποια βασικά γεγονότα. Πρώτα απ' όλα, το διεθνές δίκαιο δεν είναι άμεσα εφαρμοστέως στους ιδιωτικούς φορείς και αυτό κατά την παραδοσιακή ερμηνεία του διεθνούς δημοσίου δικαίου. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η παραδοσιακή ερμηνεία λέει ότι μόνο τα κράτη και οι δικοί τους φορείς δεσμεύονται απευθείας από διεθνείς δεσμεύσεις όπως είναι οι συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κατά τον ίδιο συλλογισμό το προσωπικό ιδιωτικών εταιριών που δεν είναι κρατικοί φορείς είτε παρέχουν είτε όχι υπηρεσίες εκ μέρους ενός κράτους δεν δεσμεύονται άμεσα από τις διεθνείς συνθήκες. Ανταυτού το παραδοσιακό εφαρμοστέο νομικό καθεστώς είναι το, τοπικό καθεστώς του κράτους στο οποίο γίνεται επιχείρηση, του λεγόμενου επιχειρησιακού κράτου. Το νομικό καθεστώς όπου δραστηριοποιείται, όπου επιχειρεί η ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλεια. Συχνά όμως έχουμε προβλήματα σε τομείς όπου υπάρχουν ένοπλες συγκρούσεις, όπου υπάρχει αστάθεια ή όπου έχουν συμβεί φυσικές καταστροφές ή όταν ε, πρόκειται για ένα κράτος παρία. Πολλές φορές δεν είναι δυνατό να υπάρξει πραγματικός έλεγχος και εποπτεία των δραστηριοτήτων ε, των εταιριών των ιδιωτικών εταιρεών παροχή ασφάλειας. Και υπάρχουν λοιπόν κάποιες προκλήσεις πολύ σημαντικέ που συνδέονται άλληλο, συνδέονται μεταξύ τους. Πρώτα απ' όλα έχουμε πολλαπλέ δικαιοδοσίε, έχουμε δυσκολίε για τη διεξαγωγή ερευνών διασυνοριακά Επίση, μεγάλο μέρο του προσωπικού δεν εμπίπτει μόνο στη δικαιοδοσία ενό επιχειρησιακού κράτου, γιατί πολλέ φορέ μετακινείται διασυνοριακά, περνάει σύνορα, ίσω περισσότερα του ενό μέσα στην ίδια ημέρα. Και επίση, δεν υπάρχει και εκπροσώπηση στην ίδια επιχειρησιακή ομάδα τη ιδιωτική υπηρεσία. Επομένω, υπάρχουν πολλαπλές ε, ε, δικαιοδοσίες ε, που μπορεί να πρέπει να εφαρμόζονται. Υπάρχει το, η εξοεδαφικότητα. Τα εθνικά επίσης νομικά συστήματα και το ποινικό δίκαιο των κρατών μελών δεν έχει συνταχθεί για να ε, αντιμετωπίζει περιπτώσεις ατόμων τα οποία κινούνται διασυνοριακά. Ιδίω πιο προβληματικό είναι όταν κάποιο διαπράξει κάποιο παράδειγμα, κάποια αξιόπινη πράξη σε μια διαφορετική χώρα. Ε, πάλι δεν υπάρχει ε, απόλυτη νομική κάλυψη. Όλες αυτές οι προκλήσεις μας οδηγούν στο τελευταίο σημείο ότι δεν υπάρχει ένα σύστημα διαφανούς λογοδοσίας για όλους αυτούς οι οποίοι παρέχουν ιδιωτικέ υπηρεσίε ασφάλειας. Αυτά τα ζητήματα, αυτές οι προκλήσεις ε, πολλές φορές ε, τα τελευταία χρόνια ήταν στα πρωτοσέλιδα, ήταν πρώτη είδηση και παρά το γεγονός ότι υπήρξαν πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, ίσως ένα γεγονός ήταν μια, μάλλον που έχετε ακούσει, είναι μια, σουηδική, μια ελβετική πρωτοβουλία Λέγονται, λέγεται το κείμενο Μοντρέ αυτό το, αυτή η πρωτοβουλία για να καθορίσει κάποιες ε, δεσμεύσεις στο πλαίσιο της ε, σύμβασης της Γενέβης. Αυτές, αυτοί οι όροι θα πρέπει να εφαρμόζονται στους ε, ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών ασφάλειας. Το Σεπτέμβριο του 2008, μετά από μελέτες, 17 κράτη συμφώνησαν και ενέκριναν το έγγραφο αυτό, το έγγραφο του Μοντρέ, που είναι ενδιαφέρουσα αντίληψη στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου σε σχέση με το, τη σημασία που έχει. Τώρα νομίζω 36 είναι τα κράτη τα οποία το έχουν προσυπογράψει. Δεύτερη πρωτοβουλία η οποία έγινε μετά από, την, ε, από το έγγραφο του Μοντρέ είναι ο Διεθνής Κώδικας Διοντολογίας ε, για τους ε, ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ICOC. Αυτό το έγγραφο επικεντρώνεται κυρίως υποχρεώσει των κρατών αλλά τώρα αφορά και τις, τους ισχυρισμούς του προσωπικού επιτόπου. Και αυτό έγινε μετά από έκκληση των ε, επιχειρήσεων, των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Παρότι είναι, ε, διέπεται από τις ανάγκες του κλάδου, είναι μια διαδικασία πολλαπλών εμπλεκομένων φορέων με στόχο να δημιουργηθούν κάποια πρότυπα που θα σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και για να υπάρξουν και μηχανισμοί ελέγχου και συμμόρφωσης. Κάποιες φορές θεωρείται αμερικανικό πρόβλημα αυτό των υπηρεσιών, των ιδιωτικών εταιριών ασφάλειας. Τα κράτη τα οποία έχουν υπογράψει τον κώδικα δεοντολογίας όμως μας δείχνουν ότι δεν είναι μόνο αμερικανικό το πρόβλημα. 43,5% των εταιριών που έχουν προσυπογράψει αυτό το έγγραφο προέρχονται από την Ευρώπη, το 24% από την Αφρική, το 21% από τη Βόρεια Αφρική και μιλώ και για καναδικές εταιρείε εδώ και βέβαια ε, υπάρχουν και κάποιες ε, εταιρείε 7 από την Ασία και μία από τη Λατινική Αμερική. 71 είναι εταιρείε που έχουν υπογράψει αυτό το έγγραφο, αλλά έχουμε και άλλε περίπου 20, οι οποίε ε, σύντομα θα ολοκληρώσουν τι διαδικασίε και θα είναι συμβαλόμενα μέλη. Οπότε θα έχουμε φτάσει σε 90 επιχειρήσει πολύ σύντομα. Τώρα, στον κώδικα διοντολογίας θα σας ε, δώσω και κάποιες συνδέσμους για να δείτε που μπορείτε να βρείτε αντίγραφα και πρέπει να σας πω ότι έχει μεταφραστεί και στα γαλλικά και γερμανικά. Ο κώδικας διοντολογίας, όπως σας είπα ουσιαστικά, θέτει κάποια ε, πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, υποχρεώσεις για την τήρηση των, και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως προβλέπεται από Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλες συμβάσεις σχετικές ε, του ΟΗΕ και αναφέρεται στις υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά ε, ε, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υποχρεώσεις που θα πρέπει να τηρούν ιδιωτικοί φορείς και επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο τώρα αυτού του κώδικα διοντολογίας τίθεται και ένα χρονοδιάγραμμα για να υπάρξει ένας φορέας ε, εποπτείας και ελέγχου ώστε να είναι αποτελεσματικός ο κώδικας διοντολογίας ε, να έχει ε, να εφαρμόζεται και να είναι αυστηρός. Και στην παράγραφο 11 του κώδικα βλέπετε μία παράγραφο η οποία ακριβώς αναφέρεται συγκρότηση ενός μηχανισμού εποπτείας και λογοδοσίας. αν δείτε τη σημερινή θα δείτε ότι τηρούνται μέχρι στιγμή, τηρείται το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει αυτό το ίδρυμα, αυτός ο θεσμός να είναι επιχειρησιακός μέχρι τον ε, Μάιο του 2012. Θα με ρωτήσετε και θα πρέπει ίσως να με ρωτήσετε τι κάνει ένας τέτοιος μηχανισμός, αυτός ο ανεξάρτητος μηχανισμός εποπτείας και συμμόρφωσης. Είμαστε στα σπάργανα ακόμα, αλλά μέχρι στιγμής έχουμε εντοπίσει τέσσερις βασικούς τομείς δράσης για αυτό το μηχανισμό. Πρώτος είναι η επαλήθευση και αξιολόγηση του κώδικα ε, δεοντολογίας μέσω ελέγχου, παρακολούθησης και πιστοποίησης. Επίσης, ε, ε, εκθέσεις και επισκοπήσεις επιτόπου, επανόρθωση, επαλήθευση σε σχέση με κάποιες καταγγελίες και βέβαια η διαχείριση του κώδικα. Τέταρτο. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες, αλλά όπως ανέφερα, εμείς συμμετέχουμε ενεργά στη δεύτερη φάση της πρωτοβουλίας αυτής. Μέχρι στιγμής μπορείτε να βρείτε πληροφορίες ε, στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Κώδικα για ε, τις ιδιωτικές υπηρεσίες www.icoc.org όπως σα είπα έχει μεταφραστεί ο κώδικας και στα γαλλικά και στα γερμανικά. Μπορείτε εκεί επίσης να βρείτε τα πρακτικά της ε, Διευθύνουσα Επιτροπής της Steering Committee βλέπετε και κάποιες συζητήσεις για το πώς πρέπει να πάρει σάρκα και οστά αυτή η πρωτοβουλία και κάποιο επιπλέον έργο. Γι' αυτό και σας παροτρύνω να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και να την ε, μελετήσετε. Τέλος, ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να σας αναφέρω κάποιες ιδέες για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε και με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή τη διαδικασία. Η πρώτη μου σύσταση θα ήταν ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση στα κράτη-μέλη για αυτή τη διαδικασία. Τα κράτη τα οποία συμμετέχουν αυτή τη στιγμή είναι η ΙΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ελβετία επίσης είναι ενδιάμεσος, ε, ένα ενδιάμεσο κράτος. Αλλά νομίζω ότι καλό θα ήταν να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή ε, περισσότερων κρατών για να προχωρήσει καλύτερα αυτή η διαδικασία. Δεύτερον, υποδητή ικανότητα ε, είστε και πελάτες και ρυθμιστές. Μπορείτε λοιπόν τα κράτη να περιλάβετε ως πελάτες πρότυπα στις συμβάσεις με τις υπηρεσίε αυτές, αλλά και ως ρυθμιστές να εφαρμόσετε ε, τις διαδικασίες και τις πολιτικές που απαιτούν συμμόρφωση. Τέλος, προανέφερα βέβαια το ίδιο, σε αυτή την επόμενη φάση που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αυτό τον μηχανισμό, επίσης μπορείτε να συμμετέχετε ενεργά τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μεγαλύτερη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτός ο διεθνής κώδικας θα μπορούσε να επιτύχει το στόχο του. Η ασφάλεια δηλαδή είτε παρέχεται από δημόσιο φορείς είτε από ιδιωτικούς να είναι πραγματικά ασφάλεια, να, παρέχει ασφάλεια για όλες και για όλους. Ευχαριστώ πολύ και περιμένω τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει ο καθηγητής κ. Ροντζίτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επειδή έχω προετοιμάσει την παρέμβασή μου στα Ιταλικά και σας έδωσα και τα σχετικά έγγραφα, θα μιλήσω στο Ιταλικά Και μετά θα απαντήσω στα αγγλικά ή στα γαλλικά στις ερωτήσεις σας. Point. I want to... Το πρώτο σημείο που θα ήθελα να σημειώσω. Θα μιλήσω λοιπόν και την ορολογία, αυτό το συμβόλαιο, τη συμφωνία θα δείχνω και τις ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας και τις ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες ασφάλειας που παίζουν όμως δύο διαφορετικούς ρόλους, έτσι. Η μία είναι εταιρεία ασφάλειας που προστατεύουν πρεσβείες σε μικρές χώρες που δεν μπορούν να έχουν την άνεση ε, να έχουν ε, φρουρούς εκεί. Έχουμε τους καραμπινιέρους ας πούμε στην ε, πρεσβεία στην Ιταλία, αλλά έχουμε μικρά κράτη που χρησιμοποιούν ιδιωτικές εταιρείες και είναι ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας. Υπάρχουν όμως και ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας στρατιωτικές, οι οποίες ε, έχουν να κάνουν πράγματα ε, σχετικά με είτε ενοπλή σύραξη είτε με σύραξη διεθνή σε το, λοιπόν σε τοπικό ή σε διεθνές επίπεδο για να τα πω όμως σύντομα εγώ θα χρησιμοποιήσω ένα ενιαίο όρο, αυτό το contractor, που θα περιγράφει και τις δύο αυτές δυνατότητες, στρατιωτική ή σχέτη ασφάλειας. Στις μελέτες μας που διεξάγουμε σε 7 πανεπιστήμια ευρωπαϊκά μαζί και το δικό μου πανεπιστήμιο στη Ρώμη. Εμείς διεξάγουμε έρευνες στα πλαίσια του 7ου προγράμματος πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ήδη έχουμε εκδώσει ένα βιβλίο σχετικά με αυτό. Αρκετές μελέτες υπάρχουν λοιπόν πάνω στο θέμα αυτό που τονίζουν το φαινόμενο της ιδιωτικοποίησης του πολέμου. Θα πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτή η ιδιωτικοποίηση του πολέμου και μέχρι ποιου σημείου μπορεί να προχωρήσει. Όπως είπε η προηγούμενη ομιλήτρια, η ασφάλεια έχει να κάνει με την απειλή κατά ενός κράτους και εάν υπάρχει χώρος και εκεί υπάρχει και όχι μόνο για τις ενοπλές δυνάμεις αλλά και τις ιδιωτικές αυτές εταιρείες. Υπάρχει κάτι το αρνητικό όμως από νομικής πλευράς, ρυθμιστικής πλευράς γιατί μας λένε αυτές οι ρυθμίσεις τι δεν πρέπει να κάνουν αυτοί οι κύριοι από αυτές τις ιδιωτικέ εταιρείε. Μια διάκριση ας πούμε ανάμεσα σε αυτούς τους κοντράκτους και τους μισθοφόρους. Τώρα τι γίνεται με τους μισθοφόρους επειδή πολλές φορές τους contractors αυτούς τους αποκαλούν ε, μισθοφόρους, άδικα επαναλαμβάνω. Αν ε, κάνουν κάτι τέτοιο, εντάξει, να τους λέμε μισθοφόρους, αλλά διαφορετικά όχι. Γι' αυτό θα πρέπει λοιπόν ε, να δούμε τι λένε ορισμένες ε, διεθνείς συμφωνίες, όπως το πρώτο προσθετικό συμπληρωματικό πρωτόκολλο της Γενέβης του 1949, το άρθρο 47, που δεν προσδιορίζει τον μισθοφόρο, αλλά λέει ότι για να είναι κανείς ε, μισθοφόρος θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από έξι στοιχεία που δύσκολα μπορεί να χαρακτηρίσουν ένα και μόνο άτομο, αλλά η δική μου άποψη είναι ότι ακριβώς ε, το χαρακτηριστικό, το βασικό είναι η συμμετοχή του η άμεση στις εχθροπραξίες. Αν δεν συμμετέχει άμεσα στις εχθροπραξίες δεν είναι μισθοφόρος. Λοιπόν, ε, έχουμε και αλλού εκτός από την ε, Σύμβαση της Γενέβης όπως για την εξάλληψη του φαινομένου αυτού ε, από την ε, Ένωση Ευρωπαϊκής Ενότητας του 1977 και επίσης του 1989 4 Δεκεμβρίου των Ηνωμένων Εθνών που απαγορεύει σε διεθνές επίπεδο τους μισθοφόρους. Θα πρέπει όμως να σκεφτούμε το εξής, ότι οι συμφωνίες αυτές δεν επικυρώθηκαν από όλα τα κρατημέλη της διεθνούς κοινότητας. Κυρίως για το πρώτο συμπληρωματικό πρωτόκολλο του 1947. Εντάξει, εκεί και τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το επικύρωσαν αλλά δεν επικυρώθηκε από τις Ηνωμένε Πολιτείες και αυτό αποτελεί από τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν στις ρυθμίσεις του εν λόγω φαινομένου. Αλλά επίσης το 1989 στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών να σας πω ότι πριν να έλθω εδώ κοίταξα να δω τι γίνεται με τις επικυρώσεις πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι 30 αλλά και όλοι επικύρωσαν, ίσως 32 κράτη και από τα ευρωπαϊκά κράτη τα 27 μόνο η Ιταλία τα επικύρωσε. Η επικύρωση είναι η μόνη χώρα λοιπόν που τη σύμβαση αυτή των Εθνών του 1989 την επικύρωσε. Βέβαια χρειάζεται κανείς να καταλάβει ότι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε είναι μεταβλητής γεωμετρίας γιατί δεν είναι στα ίδια όργανα τη διεθνή όλα τα κρατήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανήκουν. Άλλο ένα βασικό σημείο που αναφέρθηκε, θα θέλω να το επαναλάβω όμως, είναι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου προστασίας και το Διεθνές Δικαστήριο είπε όχι μόνο σε ε, συμβουλευτικές ε, εκφράσεις του αλλά και σε αποφάσεις δικαστικές ότι αυτό το δίκαιο θα πρέπει να, να εφαρμόζεται σε περίπτωση εχθροπραξιών και υπάρχει άλλο το Generalis και ο άλλο το Specialis. Ε, άλλο είναι το γενικό δίκαιο και άλλο το ειδικό δίκαιο. Αλλού ανήκει το ένα και αλλού ανήκει το άλλο. Λοιπόν, δεν θα ήθελα να θίξω τώρα αυτές τις έννοιες, να τις αναλύσω εδώ σε αυτή τη συζήτηση, αλλά και στα δύο και τα δύο αυτά θα πρέπει να εφαρμόζονται και οι δύο αυτοί κλάδοι. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και αυτό άλλωστε αποτελεί κάτι το σίγουρο, το κεκτήμενο τη στιγμή που ένα κράτος μέλος ε, έχει τον έλεγχο κάποιου κράτους ε, που δεν συμμετέχει, δεν έχει προσυπογράψει αυτή τη συμφωνία, όπως μας φάει, του Ιράκ, σε άλλη περιοχή. Ε, το κράτος μέλος όμως αυτό θα πρέπει και στο Ιράκ να σέβεται τη Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και ακόμα όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη ακόμα περισσότερο από τη στιγμή που ε, έχουμε και νομικά μέσα ε, διαθέτουμε μια ρύθμιση νομική που ενδιαφέρει τα κράτη-μέλη όταν προχωράν σε ενέργειες στο εξωτερικό. Αλλά λοιπόν όσοι αισθάνονται τον εαυτό τους θυγμένο από τον ε, κατακτητή, από τον ε, αντίπαλο, τότε μπορούν να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να ζητήσουν επανόρθωση. Ενώ το διεθνές, δεν ισχύει εδώ το διεθνές, δεν έχω το δικαίωμα βάσει του Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά πάνω σε αυτό όμως ναι, όπως είπαμε, υπάρχει δυνατότητα προσφυγής σε ενδεχόμενες ε, ενέργειες παραβίασης και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ας πούμε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Θα πρέπει να ξεχνάμε, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλα δικαστήρια που μπορούν να αποφασίσουν για μια αποζημίωση ε, που να την απαιτήσουν από εκείνον που παραβιάζει τα ανθρώπινα διεθνή δικαιώματα και νομίζω ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι όλα μέλη και της Σύμβασης της Γενέβης του 1949 αλλά και των δύο συμπληρωματικών πρωτοκόλων και σημαντικό το πρώτο πρωτόκολλο που ρυθμίζει τις με διεθνείς σειράξεις όπως ας πούμε ένα εμφύλιο πόλεμο βλέπουμε τη σημασία ενός παρομοίου φαινομένου και δεσμεύεται επίσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί πρέπει να σέβεται αυτό το διεθνέ δίκαιο και τα κράτη-μέλη θα πρέπει σε ενέργεια στο εξωτερικό να σέβονται μία εγκύκλιο που ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών το 1999 είχε ε, συντάξει για το σεβασμό αυτών των δικαιωμάτων. Εδώ για τη ρύθμιση όλων αυτών λοιπόν δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και την έννοια της άμεσης συμμετοχής της εχθροπραξίες γιατί ένα μέρος εκείνων που το μελέτησαν αυτό το φαινόμενο λένε ότι αυτές οι υπηρεσίες είναι ωφέλιμες, χρήσιμες, αλλά αυτοί οι contractors δεν θα πρέπει να συμμετέχουν άμεσα ε, στις εχθροπραξίες, γιατί τότε γίνονται κατευθυντικό, γίνονται μισθοφόροι. Και κάτι σταθερό λοιπόν το έχουμε που το επεξεργάστηκε η Διεθνής Επιτροπή επίσης του Ερυθρού Σταυρού Έχουμε όμως και παραδείγματα. Παραδείγματο χάρη, όταν έχουμε μία μεταφορά πολεμοφοδίων σε ένα χώρο και εκεί δίπλα έχουμε διεξαγωγή εχθροπραξιών εκεί ως μεταφέρει αυτές τις ε, αυτά τα πολεμοφόδια θεωρείται σαν κάποιος που συμμετέχει άμεσα στις εχθροπραξίες και αυτό δημιουργεί προβλήματα γιατί ξέρετε ότι από, το, ε, από τις υποχρεώσεις αυτών των contractors είναι και η μεταφορά Καταλαβαίνετε λοιπόν δημιουργείται πρόβλημα, παραλαμβάνω. Έχω λίγο χρόνο στη διάθεσή μου, δεν θα αναλύσω τώρα αυτό το φαινόμενο της άμεσης συμμετοχής της εχθροπραξίας, αλλά παρακαλώ προσέξτε κάτι ακόμη. Κάτι το υπάρχει στο διεθνές δίκαιο και που δεν έχουμε εξετάσει εξετάσει, δεν έχουν εξετάσει όσοι αναλύουν το φαινόμενο των contractors. Τι είναι αυτό. το έργο ατόμων που συνοδεύουν τις ένοπλες δυνάμεις χωρίς όμως να συμμετέχουν άμεσα ενεργά. Αυτά τα άτομα δεν είναι μέρος των ενόπλων δυνάμεων αλλά προσφέρουν υπηρεσίες θα πρέπει ένας από τους εμπόλεμους να τους δώσει μια σχετική άδεια και κανονικά είναι εχμάλωτοι πολέμου αν συλληφθούν αλλά η σύμβαση της Γενέβης λέει μέλη ομάδων εργασίας είτε με υπηρεσίες γιατί να βοηθήσουν έμεσα αυτές τις ένοπλες δυνάμεις. Θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας σε μια πρόσφατη έκθεση για την γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών διάβασα ότι το 54% των εργαζομένων που απασχολούνται ας πούμε στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ από τις Ηνωμένε Πολιτείε είναι contractors. Γιατί δεν είναι στρατιώτες αλλά είναι προσωπικό που κάνει πολλά και διάφορα, που προσφέρει πολλά και διάφορα σαν υπηρεσίες και δεν μπορούμε τώρα να τους εντάξουμε στο προσωπικό, στους στρατιώτες. το μαχόμενο προσωπικό. Και τώρα τι γίνεται με την πειρατεία. Ξέρουμε ότι είχαμε μία γεωμετρική πρόοδο και στο Άντεν, στον κόλπο και στον Ειδικό ωκεανό. Τι γίνεται όμως, θα πρέπει κανείς να χρησιμοποιήσει contractors για να ε, εξασφαλίσει τις ναυτικές επικοινωνίες ε, τις ναυτιλιακές επικοινωνίες ε, και τι γίνεται κοντράκτος δεν έχει τώρα για να κυνηγήσουν να πολεμήσουν τους πειρατές πέρα από το θαλασσιό Αλλά οι contractors αυτοί όμως μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υπερασπίσουν ε, πλοία από τις ε, επιθέσεις ε, των πειρατών. Αυτό δεν το βλέπουν με καλό μάτι οι διεθνείς ναυτικοί οργανισμοί, αλλά τι γίνεται, πολλά που έχουν προταθεί από την Διεθνή Ναυτιλικό Οργανισμό. Πολλά από αυτά που έχουν προταθεί μέχρι τώρα άλλα διαφορετικά δεν έχουν ε, εφαρμοστεί με επιτυχία. Τώρα για την παγκόσμια νομοθετική ρύθμιση σας είπα τι γίνεται και το διεθνές δίκαιο ε, μιλάει για το για τους ιδιωτικούς πολέμους που δεν υπάρχουν ε, ούτε οργανώσεις μισθοφόρων κανονικά. Όλες οι συμφωνίες οι διεθνείς ε, που δείχνουν τι ακριβώς συμβαίνει, τι ισχύει, όλες αυτές οι συμφωνίες ε, μιλάνε και για τις τακτικές ένοπλες δυνάμεις, εκείνους τους στρατιώτες τους ε, που πολεμούν είτε άλλοι είτε ομάδες μονάδες μισθοφόρων αλλά με στρατιωτική ρύθμιση και πειθαρχία. Άρα λοιπόν ο μαχητής ε, έχει ευρύτερη έννοια τώρα από ό,τι παλιότερα, αλλά δεν μπορεί να συμπεριλάβει τους contractors. Το 77 η σχετική σύμβαση ενοποίησε όλες αυτές τις κατηγορίες μαχητών, αλλά δεν συμπεριέλαβε τους contractors, εκτός αν συμμετέχουν άμεσα στις ένοπλες δυνάμεις, αλλά τότε αλλάζει το νόημα, αλλάζει ο όρος η έννοια. Για να δούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Η προηγούμενη εμιλήτρια είπε, δεν θα ήθελα να το επαναλάβω εγώ, εδώ για να συνοψίσω να σας πω ότι έχουμε τρία εργαλεία. Το ένα θα πρέπει ακόμα να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί. Αυτός ο Διεθνής Κώδικας Συμπεριφοράς για τους πέρχους υπηρεσιών όλα αυτά ας πούμε μετά από πρωτοβουλία της ελβετικής κυβέρνησης και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και όλα αυτά θα το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Εθνών θα διαχειρίζεται, τα συντάσσει, τα ρυθμίζει κλπ. κατά της των μισθοφόρων. Αλλά να σας πω ότι σχετικά με τους contractors πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα θα μπορούσαν όποιος και να οθήσει κανείς να συμπεριληφθούν στους μισθοφόρους ε, εδώ. Τι γίνεται με άλλες αυτές τις ρυθμίσεις. Είναι soft law αυτά, ρυθμίσεις και όχι νομοθεσία. Δεν ξέρω ποια πραγματική νομοθεσία θα ισχύσει. Εδώ η διεθνής κοινωνία είναι διαιρεμένη. Όταν έχουμε την επεξεργασία παρομοίων ε, συμβάσεων διεθνών για να μπορέσουν να εφαρμοστούν θα πρέπει όλοι να συμφωνήσουν. Δεν μπορούμε να έχουμε συμβάσεις που λίγα δυτικά κράτη μόνο τις επικυρώνουν αυτές τις συμβάσεις είτε λίγοι από τον τρίτο κόσμο θα πρέπει να διαθέτουμε εργαλεία μέσα διεθνή και να συμφωνούν όλοι πάνω σε αυτά. Και για τη σύμβαση αυτή υπάρχει μελέτη και ρύθμιση στην ομάδα εργασίας στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θεωρείται αρκετά ριζοσπαστική ο ομάδα λόγω των μελών και σχετικά με την εξακολούθηση των εργασιών της ομάδας ad hoc η... Ε, καταψήφισαν όμως οι... τα δυτικά κράτη τη συνέχιση αυτών των εργασιών αρκετά δυτικά κράτη άρα λοιπόν βρίσκει η εργασία αυτή διαιρημένους ε, τους διάφορους και τα διάφορα κράτη. Εντάξει, υπάρχει μια κάποια νομοθεσία, νομοθετική ρύθμιση, αλλά δεν ισχύει για όλους και όπως είπα στην αρχή, εμείς ε, προσπαθήσαμε να κάνουμε αναλύσεις, εξέταση νομοθεσιών διαφορών κρατών και στο ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, τα έχουμε δημοσιεύσει εκεί και σίγουρα θα έχουμε και ένα δεύτερο τόμο που θα δημοσιευθεί από ένα γνωστό εκδοτικό οίκο. Και τι είδαμε από όλα αυτά, ότι οι νομοθετικές προϋποθέσεις είναι πέρα από τις μυστικές ενέργειες στην Ιταλία ισχύει μια ιδιαίτερα απαγορευτική νομοθεσία για αυτές τις ιδιωτικέ εταιρείε ασφάλεια επιχειρήσει ε, διαχείρισης διεθνούς κρίσης. Είναι αρκετά κάμπτες ρυθμίσει, μπορούμε να το πούμε, σχετικά με αυτές ε, τις ιδιωτικές εταιρείες. Ταυτόχρονα βέβαια και για την Ιταλία, αλλά έχουν εκεί να κάνουν και να παίξουν με ένα άλλο τομέα που, όπως αυτούς ας πούμε, που προστατεύουν τράπεζες, φυλάνε τράπεζες. Θα πρέπει να δούμε και άλλα στοιχεία, άλλα θέματα ε, κατά της πειρατείας. Δεν θα πω τώρα εδώ τι έχουμε κάνει, όλα αυτά που έχουμε κάνει, αλλά έχουμε τα δύο άκρα, μια μεριά την Ιταλική νομοθεσία και από την άλλη μεριά την Βρετανική νομοθεσία. Είναι εδώ όμως εδώ ο Αρμόδιος ε, που θα μας μιλήσει για αυτά ο Βρετανός και που επιτρέπουν περισσότερα πράγματα στη Μεγάλη Βρετανία από ότι εμείς. Ε, για να ολοκληρώσω κύριε Πρόεδρε. Εκείνο όμω που εμφανίζεται καθαρά εδώ είναι ότι δεν υπάρχει μια κοινοτική νομοθεσία πάνω σε αυτό. Για ποιο λόγο. Οι ιδιωτικές εταιρείε ασφάλειας δεν υπάγονται στα πλαίσια της οδηγίας για τις υπηρεσίες του 2006 και για ιδιωτικές εταιρείε μεταφοράς και μεταφοράς χρημάτων. Θα υπάρξουν ορισμένες ρυθμίσεις, δεν έχουν υποβληθεί ακόμα όμως προτάσεις. Εγώ ε, υποστηρίζω μία πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναφερόταν εκεί ότι υπάρχει μια εντελώ ε, ε, διαφορετική νομοθεσία από το ένα κράτος στο άλλο. Θα πρέπει όμως ταυτόχρονα να αποφύγουμε αυτό το γεγονός, δηλαδή να έχουμε μια ρύθμιση, μια νομοθεσία και να υπάρχει μόνο ο ελάχιστος κοινός παρανομαστής που να εφαρμόζεται. Υπάρχουν ε, διάφορες οδηγίες ε, και διάφοροι κανονισμοί ας πούμε για την εξαγωγή αγαθών διπλής χρήσης αλλά όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν με τις σύμβασεις σχετικά με τον 428 κανονισμό του 2009 της 5ης Μαΐου του 2009 του Συμβουλίου αναφέρεται στην εξαγωγή αγαθών διπλής χρήσης και σίγουρα όσοι πάνε στο εξωτερικό και αποστέλλονται από τις εταιρείε αυτές προσφοράς παρομοίων ε, ε, ε, πρωτοβουλειών. Όσοι πάνε λοιπόν για να εκπαιδεύσουν κόσμο δεν μπορούν να χαρακτηριστούν σαν κοντράκτρος, αλλά λοιπόν δεν τους καλύπτει. Στην οδηγία 43 εδώ καλύπτεται το θέμα αυτό γιατί αναφέρεται στις διακοινωτικές διακοινωτικές εξαγωγές. Εκεί ισχύει άλλο πράγμα και υπάρχει μια ρύθμιση. Θα πρέπει να ρωτηθούμε λοιπόν εάν χρειάζεται μια κοινοτική ρύθμιση αν θα πρέπει να γίνει λοιπόν κάτι τέτοιο, κατά την αποψή μου ναι. Χρειάζεται, απαιτείται μια παρόμοια ρύθμιση και θα πρέπει να κάνουμε μία διάκριση ανάμεσα σε μια ρύθμιση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για υπηρεσίες που προσφέρονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μια ρύθμιση για υπηρεσίες που προσφέρονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όπως σας το είπα για τις υπηρεσίες, η ρύθμιση για τις εταιρείε αυτές που σίγουρα θα κάνουν και εξαγωγή αυτών των υπηρεσιών τους στο εξωτερικό. Πότε όμως θα πρέπει να υπάρξει μια κοινοτική ρύθμιση διαφορετικά θα μεταχειριστούμε αδίκως τις εταιρείε που θέλουν να εγκατασταθούν ελεύθερα κάπου θα πρέπει να δούμε και τι είναι περιοριστικό και τι είναι άλλο. Υπάρχει μια ρυθμίση εντελώ περιοριστική και μια άλλη πιο ανοιχτή, πιο φιλελεύθερη. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται, πώς να προσπαθήσουμε αυτήν τη ρύθμιση. Το κύριο μέσο εργαλείο θα μπορούσε να αποτελέσει μια οδηγία που να υιοθετηθεί ε, βάσει της τακτικής νομοθετικής διαδικασίας με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και αναφέρουμε στο 294 άρθρο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη στιγμή όμως που μία οδηγία αποτελεί ε, δύσκολο να υπάρξει, ίσως να έχουμε μια σύμφωνα και με το άρθρο 292 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής μια σύσταση που θα περιζόταν να προτείνει κατευθυντές γραμμές και μουτάτης μουτάντης κατά την απόψή μου θα μπορούσε επίσης να καταβληθεί προσπάθεια για την εξωτερική ρύθμιση προσφορές παρομοίων υπηρεσιών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 29 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ειδικά θέματα και γεωγραφικά που να είναι κάτι, ένα εργαλείο δεσμευτικό νομικά είτε και ένα soft law που να μην είναι δεσμευτικό αλλά είναι τουλάχιστον ένας κανόνας συμπεριφοράς, ένας κώδικας συμπεριφοράς που το Συμβούλιο θα μπορούσε να υιοθετήσει ε, σε μια ε, συνάντησή του και να το συμπεριλάβει σαν παράρτημα στην όλη ρυθμίση και για τον περιορισμό εξαγωγής όπλων ξεκίνησε το πράγμα από ένα κώδικα συμπεριφορά και τελικά ρυθμίστηκε το πράγμα ε, περισσότερο δεσμευτικά, νομοθετικά δεσμευτικό λοιπόν, νομικά δεσμευτικό. Κυρίε και κύριοι, ποια είναι τώρα τα συμπεράσματά μου. Τα εξής. Οι contractors είναι μιας σταθερή εικόνα ύπαρξη της σύγχρονης ασφάλειας γιατί παίζουν ρόλους σε περιπτώσεις ε, πριν, ε, κατά τη διάρκεια και μετά μια σύραξη και αρκετοί μη κυβερνητικοί οργανισμοί βρετανικοί το διαφημίζουν αυτό ότι το κάνουν ναι, όταν θα πρέπει να παίξουν ρόλο σε ιδιαίτερα δύσκολες ε, περιοχές και επίσης ε, ας πούμε για πλοία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθούν αυτές οι υπηρεσίες για να αποφευχθεί κίνδυνος πειρατείας. Κατά την απόψή μου τώρα οι βασικές προϋποθέσεις, ε, οι ελάχιστες για να μπορούν αυτές οι εταιρείες ε, να ε, εξασφαλίζουν τα εξής. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να σέβονται απολύτως τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ε, ανθρώπινο δικαίωμα. Επίσης, οι contractors δεν μπορούν άμεσα να συμμετέχουν σε μια σύραξη, σε μια μάχη. Επίσης, χρειάζεται ένας έλεγχος, ε, μια επαγρύπνηση και να δούμε ότι πραγματικά σέβονται αυτούς τους κανόνες και τέλος ε, μια ρύθμιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που απαιτείται σίγουρα και περιμένοντας ρυθμίσεις δεσμευτικές νομικά ίσως να υιοθετηθεί ένας κώδικας συμπεριφοράς ενδιάμεσα. Αυτά ολοκλήρωσα, σας ευχαριστώ, είμαι στη διάθεσή σας ή για ερωτήσεις, απαντήσεις κλπ. Merci, Σας ευχαριστώ πολύ. Ο καθηγητής ε, Μπράνοβιτς τώρα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Αγαπητέ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στο πάνελ οι ομιλητές ε, έπρεπε να κοιτάξουν κατά πόσο είναι κατάλληλο το τρέχονομικό πλαίσιο για τις δραστηριότητες των ιδιωτικών ε, εταιριών ασφάλειας και υπό ποιους όρους θα μπορούσε να είναι θεμητή και πρακτική η κρίση τους καθώς και αποτελεσματική από πλευράς ε, κόστους. Θα ήθελα να τονίσω τέσσερα σημεία τα οποία ε, έχουν να κάνουν με τον τελευταίο στόχο του πάνελ και θα ε, ήθελα να αναφερθώ σε θέματα που θα πρέπει να τα σκεφτούμε πριν αναθέσουμε τέτοιες συμβάσεις. Να ξεκινήσω με μερικές γενικές παρατηρήσεις για δύο εικασίες για το ποιο μπορεί να είναι το εύρος ε, της εξωτερικής ανάθεσης. Και μετά θα περάσω στα τέσσερα σημεία, τα οποία όλα σχετίζονται με τους συγκεκριμένους στόχους της εξωτερικής ανάθεσης και θα κλείσω την παρατηρήσή μου με κάποια σχόλια συνοπτικά σε ό,τι αφορά κάποια θέματα που ανακύπτουν από την ανάθεση τέτοιων συμβάσεων Σκεπτόμενοι την εξωτερική ανάθεση, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι γενικά ο ιδιωτικό τομέα προσαρμόζεται στι ε, ανάγκε που αλλάζουν. Άρα, ουσιαστικά είναι δυνατόν να παρέχουν ό,τι επιθυμούν οι πελάτες. Ε, οι εταιρείε μας λένε ότι, για παράδειγμα, ε, δίνουμε στις εταιρείε, στις κυβερνήσεις αυτό που επιθυμούν. Μπορούμε ακόμα και σχολεία να χτίσουμε. Άρα, τελικά, ο πελάτης αποφασίζει τι ε, δίδεται προς εξωτερική ανάθεση και τι όχι. Άρα, βάσει αυτών των ε, συμπερασμάτων θα ήθελα να εξαγάγω κάποια άλλα συμπεράσματα. Καταρχάς, προκειμένου να είναι οικονομική ε, και πρακτική η εξωτερική ανάθεση χρειάζεται, και αυτό μπορεί να φαίνεται παράδοξο, μια αναποιημένη προσέγγιση στην εξωτερική ανάθεση. Κατά δεύτερον, οι πελάτες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την ιδιότητά τους ως πελάτες σε ό,τι αφορά την εξωτερική ανάθεση. Συνήθως οι συμβάσεις αυτές ε, έχουν συγκεκριμένους στόχους και έχουν διαφορετικό περιεχόμενο. Τα τελευταία 15 χρόνια έχει αυξήσει κατά πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση την ε, δραστηριότητά της αυτής. Διάφορα προγράμματα και σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει διαφοροποιημένο σύνολο συστημάτων για το πώς μπορεί να δεσμευτεί και να ενεργήσει σε άλλες χώρες, αλλά ουσιαστικά σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικές εταιρείε ασφάλειας, τα πράγματα είναι ad hoc, δηλαδή μιλάμε για στόχους που είτε δεν έχουν προβλεφθεί, είτε για ιδιότητες που έχουν οριστεί μετα... στην εποχή μετά τον ψυχρό πόλεμο. Προκειμένου λοιπόν να είναι πρακτική αυτή η εξωτερική ανάθεση, θα πρέπει να θεωρηθεί τμήμα ενός συνολικής προσέγγισης και να ενταχθεί σε στρατηγικές ετοιμότητας. Για παράδειγμα, αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα τέλη Ιανουαρίου φέτος εκφράσει ανησυχίες για το υψηλό κόστος που προκύπτει από την εξωτερική ανάθεση σε δυτικές εταιρείε σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του προσωπικού του ε, κοινοβουλή είναι στο Αφγανιστάν και παράλληλα τονίσει ότι υπάρχουν επιτόπου ευρωπαϊκές ε, δυνάμεις ασφαλίες, ε, αστυνομία για παράδειγμα, πολιτοφυλακή, που θα μπορούσαν να κάνουν την ε, δουλειά αυτή, φαίνεται ότι θα υπήρχε δυνατότητα βελτίωσης. Άρα οποιαδήποτε ανάλυση των πόρων που χρειάζονται θα πρέπει να λάβει υπόψη τους υφιστάμενους πόρους στην κάθε χώρα μήπως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε είτε υφιστάμενου πόρους, αν, και τονίζω το αν, αν αποφασιστεί πολιτικός πώς να χρησιμοποιηθεί η αγορά, οι ιδιωτικές εταιρείες θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη σε ό,τι αφορά την εκτίμηση, εξ αρχής όμως σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των δυνάμεων. Χρειάζονται λοιπόν καλοί θεσμοί συμβάσεων δημοσίων συμβάσεων που ήδη υπάρχουν. Αυτή η ανάγκη είναι πάρα πολύ μεγάλη, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη και την πραγματικότητα που επικρατεί σε ό,τι αφορά αυτές τις εταιρείες. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι η υπόθεση οικονομικού χαρακτήρα ε, σπηλώνεται από περιστατικά απάτης ε, επιτόπου, από υψηλό πολιτικό δηλαδή και οικονομικό κόστος για παράδειγμα τις κατηγορίες σεξουαλικής εμπορίας στη Βοσνία, στο ε, KBR στα πρώτα ε, χρόνια της ε, εισβολής στο Ιράκ. Αν θέλουμε η εξωτερική ανάθεση να είναι επιτυχής, θα πρέπει να συμμετέχει ενεργά η εταιρεία. Τι σημαίνει όμως αυτό. Οι ΙΠΑ μας διδάσκουν με τις επιτυχίες και τις αποτυχίες τους σε μια πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύθηκε πριν από δύο, χρόνια, πριν από δύο εβδομάδες αναφορικά με το Αφγανιστάν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έκανε κάποιες συστάσεις ε, για το πώς καταρχάς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα φτωχά αποτελέσματα της εξωτερικής ανάθεσης και, μπορούμε, και πώς μπορούμε να θεσμοθετήσουμε μακροπρόθεσμα κάποιες αλλαγές. Τέσσερα σημεία φαίνεται ότι είναι πιο σημαντικά από τις συστάσεις αυτές. Καταρχάς ότι θα πρέπει να υπάρχει ομογενοποίηση των ε, Πολύ συχνά παρέχονται οι ίδιες υπηρεσίες από διάφορες εταιρείες, από διάφορα ε, όργανα. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά προγράμματα ΚΕΠΑ, υπάρχουν πολλές δράσεις ε, κρατών μελών στην ίδια χώρα. Θα πρέπει να υπάρχει μια ενοποίηση των απαιτήσεων. Αυτό βελτιώνει και τις απαιτήσει, αλλά βελτιώνει και το κόστος. Επίσης, συντονισμένες και ακριβώς ορισμένες ανάγκες σε μια κατάσταση όπου επικρατεί ανταγωνισμός από πλευρά προμηθευτών. Άρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και αυτή την έννοια του ανταγωνισμού. Το σύστημα το αμερικανικό είναι καλό για την ομογενοποίηση των αναγκών σε φάση σχεδιασμού πριν από την ανάπτυξη των δυνάμεων, αλλά θα πρέπει να διατηρηθούν και κάποιες δυνατότητες εξόδου και η δυνατότητα να στραφεί κανείς σε κάποιον ανταγωνιστή. Άρα χρειάζονται κάποιες πληροφορίες για την μηχανική βάση και για τη βελτίωση ενδεχομένω των συμβατικών όρων. Ένα άλλο θέμα έχει να κάνει με το πώς μπορούμε να ελέγχουμε ε, τι εταιρείε αυτές επί τόπου. Χρειάζονται λοιπόν ε, λογοδεσία. Σε περιπτώσεις και υποθέσεις ε, όπου επικρατούν προβλήματα στη χώρα που αναπτύσσονται οι δυνάμεις, είναι θέμα του πελάτη να καλύψει αυτό το κενό και ένας τρόπος είναι να αναπτυχθεί μια δύναμη επιτόπου που θα γνωρίσει τις ανάγκες ε, της περιοχής. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας τρόπος για να μειωθεί το κόστος και έτσι μπορεί να συμβάλλει στην αξιολόγηση ε, δεδομένων ε, προηγουμένων αποστολών. Και από αυτή την άποψη η βασική ε, ο βασικός όρος για μια καλή ανάλυση του κόστους είναι να υπάρχει από πλευράς του πελάτη μια καλή αντίληψη του κόστους για την ε, εκπαίδευση του προσωπικού. Άρα το βασικό ερώτημα είναι πώς το πετυχαίνουμε αυτό και εδώ απαντώ αναπτύσσοντας ε, μια συντονισμένη στρατηγική βάση πέντε σημείων κίνησης. Καταρχάς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις συμβάσεις αυτές ως ε, μια κεντρική λειτουργία μέρος του συνολικού, της συνολικής αποστολής. Δεύτερον, θα πρέπει να δημιουργηθούν γραφεία συντονισμού σε επίπεδο συμβάλλοντα και να υπάρχουν σαφές, αρμοδιότητε. σαφές αρμοδιότητες τα γραφεία αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως διεπαφές για τον καλύτερο συντονισμό. Μπορούν να ελέγχουν την καλή εφαρμογή των συμβάσεων και όπου είναι απαραίτητο να ξεκινήσουν κάποιες αλλαγές ε, στη σύμβαση. Για να επιτευχθούν αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να προταθούν ε, να προταθεί μία να προταθούν απαιτήσει ε, πιστοποίησης και εκπαίδευσης του προσωπικού κατά τέταρτον παρά το γεγονός ότι μάλλον οι έρευνες καταδεικνύουν ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος σε περίπτωση που δεν είναι οικονομικές αυτές οι συμβάσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ε, λόγος να υπάρχει τέτοια εξωτερική ανάθεση, ιδιαίτερα όταν η πόρη είναι πληρισμένη. Αν υπάρχει χρόνος να υπάρχουν συγκεκριμένες συμβάσεις και τέλος, να δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων με τους ε, παρόχους των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Αυτή η βάση δεδομένων spot, όπως αναφέρεται, χρησιμοποιείται στις είπε και μπορούσε, θα μπορούσε να αποτελέσει υπόδειγμα για το πώς θα λειτουργούσε μια ευρωπαϊκή τέτοια βάση δεδομένων. Ένα γενικό θέμα τώρα για το πώς ε, χρησιμοποιούμε τις ε, ιδιωτικές εταιρείες στρατιωτικής ασφάλειας. Μισό λεπτό. Τα πιο πολλά αρνητικά αποτελέσματα αποτελούν προσωρινά προβλήματα. Άρα, όσο πιο μεγάλο είναι το χρονικό διάστημα κατά το οποίο υπολογίζουμε υπολογίζουμε σε τέτοιε εταιρείε, τόσο πιο περιορισμένο είναι ο κίνδυνο για εγκληματικέ δραστηριότητε, για αρνητικές συνέπειες. Γιατί οι εταιρείε αυτέ ε, γνωρίζουν έτσι το περιβάλλον και εντοπίζουν ποιες δραστηριότητες είναι παράνομες. Αυτό αποτελεί μια παρατήρηση κάποιων υπηρεσιών μόνον. Και δεν θέλω να πω ότι είναι ένα, μια σίγουρη διαπίστωση. Ωστόσο, ένας τρόπος για να περιορίσουμε τους κινδύνους της εξωτερικής ανάθεσης και να πετύχουμε μια οικονομική ανάθεση είναι να παρατηρήσουμε τι γίνεται κατά την εφαρμογή των συμβάσεων. Οι στρατηγικές θα πρέπει να έχουν ως στόχο να μεταφέρουν αυτές τις δυνατότητες σε δημόσια ικανότητα. Για παράδειγμα, η αρχή εκπαίδευσης των εκπαιδευτών, η οποία ήδη εφαρμόζεται στο Αφγανιστάν. Είναι μια, ένα καλό παράδειγμα για το πώς μια βιώσιμη προσέγγιση μπορεί να λειτουργήσει και για το πώς η ανάθεση στρατιωτικών ε, επιχειρήσεων στρατιωτική ε, εκπαίδευση μπορεί να λειτουργήσει. Η ιδέα είναι απλή και αποτελεσματική. Ξεκινάμε να εκπαιδεύουμε με 10 σημασιούχου που ε, εκπαιδεύουν για παράδειγμα μία αστυνομική μονάδα αλλά παράλληλα εκπαιδεύονται και μονομένοι αστυνομικοί προκειμένου να εκπαιδεύσουν αυτοί στο μέλλον. Περιορίζουμε, περιορίζουμε έτσι τα ιδιωτικά μέσα χρησιμοποιώντας δημόσιους πόρους για την εκπαίδευση. Όσο δύσκολες και αν είναι αυτές οι αρνητικές συνέπειες, είναι προφανώς κοιτώντα τις επιχειρήσεις, μάλλον τις απόπειρες ε, που γίνονται στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, να αποκλείσουν ε, αλλοδαπές τέτοιες εταιρείες, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι υπάρχουν πιο πολλά προβλήματα με τις εγχώριες εταιρείε. Υπάρχουν από στρατηγικές ε, πολύ καλοί λόγοι για να χρησιμοποιηθούν εσωτερικές εγχώριες εταιρείε, γιατί, για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη γνώση των εταιρεών αυτών ε, για την περιφέρεια, την περιοχή. Επίσης, ε, μπορεί να έχουν δικαιοδοσία. Ένα άλλο επιχείρημα για την υπέρ της χρήσης ε, ιδιωτικών εταιριών είναι ότι η εταιρεία με τον τρόπο, η αγορά με τον τρόπο αυτό μπορεί να απορροφήσει τους ανειδίκευτους, ε, τα ανειδίκευτα άτομα τα οποία που συμμετείχαν σε τέως παραθεωρητικές οργανώσεις, οι ένοπλες ομάδες μπορεί να μετατρέψουν ε, τους πρώην αντάρτες σε ε, άτομα τα οποία νόμιμα εργάζονται σε τέτοιες ιδιωτικές εταιρείε. και αυτό μπορεί να βελτιώσει τις δυνατότητες και την ικανότητα των ε, αποστολών ιδιωτικής ασφάλειας για να το θέσω διαφορετικά, η χρήση τους από την διεθνή κοινότητα δεν θα ήταν αποτελεσματική από πολιτικής άποψης, αλλά δεν είναι μόνο οι μη κρατικοί φορείς εκείνοι που υποφελούνται από την ιδιωτική αυτή διάσταση της ασφάλειας. Για παράδειγμα, στην Αγγόλα, πολλές τέτοιες εταιρείε απασχολούνται από κυβερνητικούς αξιωματούχους. Αυτή η βρυδική υπόσταση δεν εμπλέκεται και δεν συμβάλλει στην οικοδόμηση κρατικών θεσμών. Αλλά τέλος, πολλές ε, τέτοιες ομάδες εξακολουθούν να διαθέτουν μικρά όπλα και άρα δεν προχωρά η διαδικασία για τα προγράμματα τα οποία αποκαλούνται DDR για αφοπλισμό, αποστράτευση και επανένταξη. Άρα, δεδομένων όλων αυτών, η χρήση της ιδιωτικής αγοράς των ιδιωτικών εταιριών ασφάλειας από την διεθνή κοινότητα συμπεριλαμβάνει και πολλούς κινδύνους σε ό,τι αφορά την ε, αντιμετώπιση κινδύνων. Θα ήθελα συνοψίζοντας να κλείσω και να αναφέρω κάποια συμπεράσματα. Όπως μας δείχνει το παράδειγμα των ΗΠΑ, κάποιες ε, χώρες, οι χώρες μάλλον που εξετάσουν την εξωτερική ανάθεση θα έπρεπε να κοιτάξουν να εφαρμόσουν κατάλληλα μέτρα προτού καταλήξουν να εξαρτώνται υπερβολικά από τέτοιες εταιρείε και να καταλήξουν σε ένα αδιέξοδο όπου ουσιαστικά δεν μπορούν να αποσύρουν αποφάσεις εξωτερικής ανάθεσης. Άρα κατά συνέπεια, αν, τονίζω πάλι το αν, αν πολιτικά αποφασιστεί να γίνουν εξωτερικές αναθέσεις θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να ξεκινήσει μια ρεαλιστική προσέγγιση και να γίνει επένδυση στις δυνατότητες ελέγχου της όλης διαδικασίας. Πέρα από αυτό το εσωτερικό στοιχείο περί των οργανώσεων, ένα βασικό θέμα το οποίο θα πρέπει να προωθεί είναι η ε, ρύθμιση. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε την ε, ευθύνη που προκύπτει από την ρύθμιση, αλλά και το πολιτικό όφελος. Για παράδειγμα, ο Διεθνής Κώδικας Διαντολογίας μπορεί να συμβάλλουν σε μια εξορθολογισμό της βιομηχανίας του κλάδου, ε, θέτοντας υψηλά πρότυπα. Ο θετικός ε, αντίκτυπος για τους πελάτες είναι ότι ουσιαστικά οι αδύναμες εταιρείε δεν επιβιώνουν. Άρα το βασικό μήνυμα είναι το εξής. Αν θέλει κανείς το outsourcing, την εξωτερική ανάθεση και δεν το λέω αυτό επειδή το υποστηρίζω, απλά εννοώ ότι αν θέλουμε να αποδώσει οικονομικά η εξωτερική ανάθεση, είτε οικονομικά είτε πολιτικά, θα πρέπει να επενδύσουμε σε τέτοιες οργανωτικές δυνατότητες εκ των προτέρων. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Και τώρα θα παρεύουν οι συνάδελφοι, όσοι το επιθυμούν. Κύριε Λεζή, με ζήτησε το λόγο. ευχαριστώ πολύ äh, για τις ε, παρεμβάσεις σα και για την εισήγησή σας. Κάποια γενικά στοιχεία. Νομίζω ότι το κρατικό μονοπόλιο στη βία έχει ένα νόημα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του πολιτισμού θα πρέπει να πω παράλληλα ότι και το κρατικό βία δυστυχώ δεν αποτελεί καμία ασφάλεια για τις παρεμβάσεις. Και εδώ πέρα φαίνεται ιδιαίτερα πόσο καλό παράδειγμα είναι η φρεχτή ιστορία της χώρας μου. Όταν προετοιμάστηκα για το πάνελ αυτό, είχα την αίσθηση ότι χανόμουν σε μία ζούγκλα, γιατί πραγματικά και η προσφορά των ιδιωτικών αυτών ε, εταιριών είναι τόσο μεγάλη και ποικιλόμορφη που δεν είναι εύκολο να βρει κανείς μία ενιαία γραμμή. Κατά δεύτερον, πρώτες εντυπώσεις θα ήθελα να πω ότι και η δικτύωση των υπηρεσιών αυτών, ποιος παρέχει ποιες υπηρεσίες και ποιος αναθέτει ποιες υπηρεσίες σε ποιον. Και τι ακριβώς αναθέτει για αναθέτει θέματα ασφαλείας, πρόκειται για πετρελαϊκές εταιρείε που θέλουν να εξασφαλίσουν την ασφάλειά τους. Είναι δημόσιες τέτοιες επιχειρήσεις, υπάρχουν και μυστικές τέτοιες αναθέσεις. Τι προσφέρουν αυτοί οι πάροχοι. Μιλάμε για στρατιωτικές και ε, αποστολές. Μιλάμε για παροχή όπλων σε περιοχές κρίσης και μόνο και μόνο λοιπόν αυτή η διαπλοκή και η πολυμορφία των υπηρεσιών αυτό με μπερδεύει. Δεν μας επιτρέπει να ξαδιαλύνουμε τα πράγματα. Και εδώ έχω να ρωτήσω το εξής. Νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λόγος το ότι διοργανώνουμε εδώ αυτή την ακρόαση. Υπάρχει λόγος και νομίζω ότι αυτό μας, μας απασχολεί δεν είναι μόνο η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, αλλά και η εφαρμογή του κράτους δικαίου, η εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άρα διερωτώμε σε ένα τόσο πολυσύνθετο περιβάλλον, όσο και αν υπάρχουν δυνατότητες και πραγματικά ε, θεωρώ ότι αξίζει να το σκεφτούμε. Αξίζει να σκεφτούμε και την ανάπτυξη ενός κώδικα διοντολογίας. Να διαρωτώμε όμως τι δυνατότητα υπάρχει να καταστεί δεσμευτικό ένα τέτοιο κώδικα. Για παράδειγμα, μια παράνομη κυβέρνηση, ένας παράνομος κυρίαρχος, ένα αποτυχμένο κράτος το οποίο εμπλέκεται με, σε έναν εμφύλιο πόλεμο με διάφορες οργανώσεις ένας τέτοιος ε, φορέας λοιπόν αναθέτει σε μισθοφόρους και σε μια οργάνωση μισθοφόρων ε, που εμπλέκει μισθοφόρους από όλον τον κόσμο. Ε, ωραία, έστω ότι υπάρχει ο κώδικας. Ποιος θα είναι ο κατηγορούμενος όταν θα διαπιστωθούν παραβιάσεις του κώδικα αυτού, όταν δεν υπάρχει νομική βάση για την ανάθεση της σύμβασης. Αυτό λοιπόν διαρωτώμε πώς σε μια τόσο πολύ κατάσταση είναι δυνατόν να αναπτυχθεί οποιοδήποτε δεσμευτικό κανόνας. Και κατά δεύτερον, να θέσω μια γενικότερη ερώτηση. Μέσω πρόθεσμα, μακρύ πρόθεσμα και από βιώσιμη πλευράς, ποια είναι η επιρροή της εξωτερικής αυτής ανάθεσης σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη κρατικών δομών. Ποια είναι η επιρροή, πώς επηρεάζει η ανάπτυξη στρατιωτικής βίας, την ανάπτυξη κρατικών δομών σε όλο τον κόσμο και μήπως αυτό συμβάλλει σε αυτό που πάντα κατηγορεί τον εαυτό της η Ευρωπαϊκή Ένωση, την ε, δημιουργία αποτυχημένων κρατών. Αυτή η μισθοφόρη, αυτή η ανάθεση του κρατικού μονοπωλίου μακροπρόθεσμα δεν οδηγεί σε μια πολυμορφία των ε, οργανώσεων αυτών και σε μια διάλυση των κρατικών δομών. Να παρατηρήσω επίσης ότι είναι τελείως διαφορετικά τα συμφέροντα σε ό,τι αφορά τη, τους πολέμους. Ένα μικρό παράδειγμα. Ο κόσμος τι θέλει. Θέλει να τελειώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται ο πόλεμος. Μία εταιρεία η οποία ωφελείται από τον, επωφελείται από τον πόλεμο αυτό, λογικό είναι ότι έχει συμφέρον να διονυστεί όσο το δυνατόν γίνεται ο πόλεμος αυτός. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι δυνατόν να το υποστηρίξουμε. Και αυτό θεωρώ ότι δεν θα αντιμετωπιστεί με τη θέσπιση ενός κώδικα δεοντολογίας. Ευχαριστούμε. Αναγκόμες τώρα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσουμε για την τόσο σημαντική ενδιαφέρουσα αυτή πρωτοβουλία και ακούγοντας ε, τους τρεις πρώτους αυτή τη γνώμη σχημάτισα, το ίδιο θα γίνει και στη συνέχεια. Είναι πήγον ε, εδώ το Κοινοβούλιο να βοηθήσει όλα αυτά και να ενεργήσει ταυτόχρονα, να δραστηριοποιηθεί με συγκεκριμένες συστάσεις στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Η συνάδελφος Λέζιν μίλησε για ζούγκλα. ζούγκλα και ένας ε, Αμερικανός ε, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνομιλώντας με εκείνον μου είπε ότι είναι πιο εύκολο να λειτουργήσει ένα τσίρκο στις ε, Ηνωμένε Πολιτείες. παρά μια εταιρεία ε, ε, ιδιωτική ασφάλειας. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν όλα αυτά. Και εδώ αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση που είναι ανάλογη των όσων ισχύουν στο οικονομικό επίπεδο σε διεθνές, σε, στο διεθνή χώρο. Ε, πριν τα πράγματα ήταν καταβούληση και τώρα προσπάθ, γίνεται προσπάθεια να υπάρξει μια ρύθμιση. Ε, ίσως είναι αργά όμως, δεν πρέπει να χάσουμε σαν κοινοβούλιο εμείς χρόνο και υποβάλλω μια πρόταση να συσταθεί μια, μάλλον να υπάρξει μια έκθεση με τις ε, σχετικές συστάσεις συγκεκριμένε στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο και ξέρω ότι στα πλαίσια αυτά τα πανεπιστημιακά έχει γίνει ήδη πολύ καλή δουλειά όπως και στον ΟΗΕ στη Γενέβη μαζί και με τα όσα ακούσαμε και θα ακούσουμε σήμερα από τους εμπεριγνώμονες εδώ. Και πολύ σημαντικό είναι επίσης να ακούσουμε και την ίδια τη βιομηχανία. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τους εμπειρογνώμονές μας πίσω συγκεκριμένα παραδείγματα γιατί ε, αργότερα με τους ε, για να δούμε και με τους με τους ε, υπαλλήλους του Συμβουλίου, μήπως εσείς θα μπορούσατε να μας δώσετε παραδείγματα. Τι γίνεται για, και για την εξωτερική πολιτική γενικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι γίνεται ε, ε, μπροστά σε ένα παρόμοιο κίνδυνο, σε παρόμοιο δίλημα, τι μπορούμε να κάνουμε. Ο τελευταίος ομιλητής ε, μίλησε, ο κύριος Μπράνοβιτς, μας έδωσε ένα παράδειγμα με την Γερμανία που έκλεισε μια συμφωνία με κάποιον για να είναι σύμβουλος και επίσης για τους εκπαιδευτές του Αφγανιστάν. Θα πρέπει να δούμε μια συντορισμένη πολιτική ελέγχου και προσλήψεων και καλό θα ήταν να έχουμε και άλλα συγκεκριμένα παραδείγματα. Εντάξει, δεν μιλάω μιλάω γενικά για την εξωτερική πολιτική. Για να πάρουμε το παράδειγμα τώρα του Ιράκ υπηρεσίες ασφάλειας σε όσους μας εκπροσωπούν στην αντιπροσωπεία πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιος προστατεύει και επίσης ε, αποστολές ε, προεκλογικής ε, παρουσίας, παρατήρησης. Τι γίνεται. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτές τις εταιρείες λοιπόν. Θα ήθελα συγκεκριμένα παραδείγματα, αν όχι σήμερα, τουλάχιστον ε, μια κάποια άλλη στιγμή. Μήπως θα μπορούσατε να μας δώσετε αυτές τις πληροφορίες και κάτι ακόμα. Είναι πολύ σπουδαίο να σκεφτόμαστε κάτι που αναφέρθηκε σχετικά με τις ε, υποχρεώσεις μας ε, στα πλαίσια με αποστολές ας πούμε από τη στιγμή που τραβούν σε μακροσυράξεις γιατί θα πρέπει ίσως να δούμε μήπως έχουν ε, σίγουρα ε, ένα ε, συμφέρον να παραταθούν αυτές οι κρίσεις από πλευρά των εταιριών είτε σχετικά με τα όπλα κλπ. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα για να μπορέσουμε να συντάξουμε και τις συστάσεις μας. Ευχαριστώ. Ρομπέρτο, εδώ γρήγορα γρήγορα έχουμε τους τρεις ομιλητές ε, που θα πρέπει να έχουμε που θα πρέπει να έχουν χρόνο. Μήπως μπορείτε να τα πείτε γρήγορα γρήγορα κι εσείς. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και την Αναγκόμες. Είπε αρκετά από αυτά που ήθελα να πω εγώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές μας για όλα αυτά τα ιδιαίτερα χρήσιμα που μας είπαν πάνω σε μια πραγματικότητα που ισχύει. Θα πρέπει να υπάρξει ρύθμιση εκεί είναι ζούγκλα αυτή σχετικά με το διεθνές δίκαιο. Θα ήθελα να υποβάλω δύο-τρία συγκεκριμένα ερωτήματα. Εντάξει, δεν θα επανέλθω για την ανάγκη ε, σύσταση από πλευρά Κοινοβουλίου, όπως το είπε ακριβώ και ο καθηγητής Ροντζίτη, είναι κάτι το πολύ σημαντικό και υπάρχει μια δυσκολία να πετύχουμε ένα πλαίσιο νομοθετικό με τους κύριους πρωταγωνιστές με γενικό τρόπο και γι' αυτό χρειάζεται μια πρωτοβουλία ακόμα περισσότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο για αυτή τη ρύθμιση. Αλλά για τον καθηγητή Ροντζίτη θα ήθελα να ρωτήσω το εξής από νομικής πλευράς μίλησε και σωστά στο δεσμευτικό, για το δεσμευτικό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για ενέργειες πέρα από το χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν ρίξουμε όμως μια μάτια στο πλαίσιο της συνθήκης Λισαβόνας, τι γίνεται πέρα από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το εσωτερικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι δεσμευτικά νομικά σχετικά με το χώρο ασφάλειας, δικαιοσύνης κλπ. σχετικά με τις εξωτερικές ενέργειες και επιχειρήσεις και δεν υπερισχύει και του διεθνούς δικαίου σχετικά με παρόμοιες αποστολές. Θα πρέπει να δούμε τη Λισαβόνα. Δεν ε, προσδιορίζει ακριβώ αυτό το εσωτερικό δίκαιο. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται, γιατί δημιουργεί ένα πρόβλημα στι αποστολέ μα στο εξωτερικό, νομική ε, υφή ε, και νομίζω ότι θα ενδιαφέρει όσου όλου ασχολούνται, εργάζονται πάνω σε αυτό. Και επίση για τον Μπράνοβιτ να ρωτήσω κάτι. Περισσότερε διευκρινήσει, δηλαδή εδώ στο Κοινοβούλιο νομίζουμε ότι οι contractors δεν χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά, τουλάχιστον σχετικά με το κόστος όφελος σε μας επιχειρήσεις όπως το Ιράκ, στο Αφγανισμό. Και βλέπουμε ότι είναι αυτά τη στιγμή που πρέπει να πληρώσουμε το λογαριασμό και βλέπουμε το ιδιαίτερα υψηλό κόστος. Υπάρχουν μελέτες από πλευράς του Πανεπιστημίου σχετικά με αυτό το κόστος όφελος. Θα θέλαμε ακριβώς να έχουμε μια καλύτερη επαφή με την Επιτροπή αυτή για τα εξωτερικά θέματα θέματα και θα θέλαμε να ακούσουμε και τη δική σας άποψη ε, εκτός όλων αυτών να μας πείτε πώς τα βλέπετε. Τελευταίος, τελευταίος Γρήγορα γρήγορα. Ο Αλήν εκπρόσωπος. Πρόεδρε, ε, αναφυσβήτητα αυτό που συζητάμε σήμερα είναι μια πραγματικότητα. Και σίγουρα δεν αρκεί απλώς να την εξορκίσουμε ούτε να κάνουμε ότι δεν υπάρχει. Δεύτερο συμπέρασμα, χρειάζεται ρύθμιση. Γιατί το περιβάλλον είναι απόλυτα απορριθμισμένο δεν έχουμε μια σαφή εικόνα τι γίνεται, πώς γίνεται, κατά ποιους κανόνες γίνεται. Εγείρονται εξάλλου και άλλα θέματα σημαντικά. Αγγίζει τον πυρήνα της εθνικής κυριαρχίας. Έως τώρα ξέραμε ότι τα θέματα ασφάλειας ήταν στον πυρήνα της εθνικής κυριαρχίας. Μπορούμε να εκχωρήσουμε τόσο σημαντικό τμήμα της εθνικής κυριαρχίας σε ιδιωτικές εταιρείε. Είναι ένα μεγάλο πολιτικό πρόβλημα αυτό. Παραδείγματο χάρη υπάρχουν και άλλα επιπλέον προβλήματα εάν σε ένα failed state γίνεται μια μίσθωση με εταιρεία ιδιωτική ασφαλείας και ακριβώς επειδή είναι failed state μετά από λίγο δεν έχει να πληρώσει την εταιρεία αυτή. Αυτοί οι άνθρωποι τι θα κάνουν. Δεν έχουν την πίστη, την εθνική ή τη δέσμευση απέναντι στο κράτος τους. Είναι απλώς μια ιδιωτική εταιρεία. Πώς θα καλύψουν τα συμφέροντά τους. Πώς θα αναζητήσουν τα χρήματα που δεν θα παίρνουν. Μπορεί να οδηγήσουν σε καταστάσεις πολύ δύσκολες. Δύο ερωτήσει. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ κρατών και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Εάν κράτη προχωρούν σε συμβόλαια με τέτοιε εταιρείε, αυτά τα συμβόλαια δεν θα πρέπει να αποδώσουν αποτελέσματα ή να εγκριθούν εάν δεν υπάρχει προηγούμενη έγκρισή του από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Δηλαδή ένα κράτο που θέλει να κάνει ένα συμβόλαιο αυτό το συμβόλαιο θα πρέπει να πηγαίνει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και μόνο αν υπάρξει απόφαση σύμφωνη γνώμη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και κάτω από διάφορα κριτήρια θα μπορεί να γίνεται ένα συμβόλαιο. Είναι μια σκέψη. Τώρα όσον αφορά τις ιδιωτικές εταιρείες που μισθώνουν ε, ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας, εκεί υπάρχουν πολλά ζητήματα. Πάρτε το παράδειγμα της πειρατείας. Μπορεί μια ναυτιλιακή εταιρεία να μισθώσει και να βάλει στα καράβια της μια ιδιωτική εταιρεία ασφάλειας ποιοι θα είναι οι κανονισμοί εμπλοκής, τα rules of engagement. Ποιος ξεκινάει πρώτος να κάνει τι. Εγείρονται λοιπόν μια σειρά από και είμαι βέβαιος ότι οι εμπειρογνώμονε που είναι εδώ παρόντες θα μπορέσουν να μας διαφωτίσουν σε εμά που είμαστε αδαείς και για πρώτη φορά ασχολούμαστε με το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Τρία με τέσσερα λεπτά ο καθένας. Καθηγητά κύριε Ροντσίτη, έχετε το λόγο πρώτος. Thank you, thank you very much, Mr. President. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για το πρόβλημα της ευθύνης που ήταν το πρώτο ερώτημα που μου τέθηκε. Πιανού ευθύνη είναι. Είναι δύσκολο να το απαντήσουμε το ερώτημα αυτό, αλλά καταρχήν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ευθύνη του κράτους έδρας, host state, αλλά και του κράτους που απασχολεί αυτές τις δυτικές εταιρείες. ένας, έχουμε το κράτος Χ το οποίο έχει, το, στο οποίο έχει την έδρα του μια ιδιωτική εταιρεία και το κράτος Ψ που είναι το κράτος στο οποίο ασκεί τη δραστηριότητά του. Και οι δύο είναι υπεύθυνοι. Και οι δύο χώρες είναι υπεύθυνοι. Τώρα όταν μια εταιρεία ε, είναι κάπου καταγεγραμμένη, εγγεγραμμένη, ε, σαν να έχει μια σημαία ας πούμε ευκαιρία. πάλι ε, Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να ισχύει και για τους ε, ανάδοχους αυτούς, τους contractors. Είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν, κάποιες φορές υπάρχει σύγχυση και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε ποιο είναι το υπεύθυνο κράτος σε κάθε περίπτωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το συμβόλαιο, να δούμε κατά πόσον τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι διεθνείς συνθήκες, στο ανθρωπιστικό δίκαιο. Ναι, μπορούμε να βάλουμε όρους στα συμβόλαια, αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη μα ότι αυτά τα προβλήματα ασφάλεια, αυτές οι ανησυχίε είναι πολύ πραγματικές και είναι πολύ δύσκολο να επεξεργαστούμε μια πολιτική όπου οι εταιρείε θα πρέπει να εκδίδουν κάποιο συμβόλαιο. of international crimes. Αν θέλουμε να προσαγάγουμε στη δικαιοσύνη αυτούς που έχουν διαπράξει αξιόπινες πράξεις, έχουμε ε, διάφορες διατάξεις, σόφα παραδείγματος χάρη, και έχουμε δει παραδείγματα όπως ε, στο Ιράν, έχουμε δει τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, αλλά υπήρχαν αρχικά και κάποιες ιδιωτικές εταιρείες οι οποίοι είχαν καθεστώς ατιμορρησίας, ασυλίας και δεν μπορούσαν να διωχθούν από κράτη. Αυτό πρέπει να το πούμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δεύτερη παρέμβαση, συμφωνώ πλήρως και είπα ότι κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. έχουμε και κάποιες αποστολές. Παραδείγματο χάρη στο Ιράκ. Ή ε, αποστολές εκλογικής παρατήρησης. Ενδέχεται να χρειαστούν προστασία αποστολές αυτές. Άρα πρέπει κάτι να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά πρέπει να έχουμε μια ρεαλιστική προσέγγιση. Κυρία μου, μιλήσατε για το πρόβλημα της διάδοσης όπλων από τις εταιρείες αυτές. Στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπάρχει ένα σχέδιο εγγράφου το οποίο ε, έχει συνταχθεί και αν θυμάμαι καλά υπήρχε μια διάταξη κατά του ε, όποιου χρησιμοποιεί ε, πυρηνικά όπλα και ήταν απίστευτο επειδή ήρθαν και μα ζήτησαν συμβουλή, εγώ έγραψα σε αυτού. και το μα είναι δυνατόν να μιλάμε για χρήση, μάλλον χημικών όπλων. Μπορεί να χρησιμοποιήσει κανεί χημικό όπλο. Εντάξει, είναι εύκολο να τα φτιάξει κανεί, αλλά το να τα χρησιμοποιήσουμε είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, διαγράψτε αυτή τη ρήτρα για τα χημικά όπλα του είπα. Είναι πραγματικά άνευ νοήματος. Και είναι ένα θέμα οικουμενικό. Είναι το θέμα της οικουμενικότητας, οικουμενικής ισχύω των συμβάσεων αυτών. Μπορεί να βάλουμε όλες αυτές τις ωραίες ρήτρε, αλλά τα άλλα κράτη να μην ε, επικυρώσουν ε, την ε, σύμβαση. Άρα θα είναι τελείως ανευνοήματος η όλη προσπάθεια. Ο κύριος Γκουαλτιέρη τώρα. Πολύ σωστά τα είπε. Πρέπει να δούμε ακριβώ την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων, αλλά και τη συνθήκη και το κεφάλαιο, τη χάρτα που είναι προσαρτημένη σε αυτό και το κεφάλαιο 6, το άρθρο 6. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση προβλέπει τη δυνατότητα αναστολή τη ισχύω τη σύμβαση. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Υπάρχει σκηνοποίηση στο Γενικό Γραμματέα ότι δεν πρόκειται να εφαρμοστεί η ε, σύμβαση. Που μπορεί κάποιο να, να την κάνει αυτή την κοινοποίηση. και τηρεί πλέον μόνο τις ρήτρε ε, που ε, αφορούν κάποια ελάχιστα, κάποια κατώτατα κατώτατες υποχρεώσεις, παραδείγματο χάρη ε, αποφυγή βασανισμών κτλ. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Όταν μιλάω για την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ποιο είναι το πρόβλημα. Έχουμε ενδικά μέσα εδώ κατά του κράτου που ε, είναι δύναμη κατοχή σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Στο Στρασβούργο μπορεί κανείς να προσφύγει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων. Έχω πει και το επισήμανα πριν είναι πάρα πολύ σημαντική η ποινική δικαιοδοσία. Αλλά πολύ σημαντικό είναι και το ένδικο μέσο που υπάρχει για να υπάρξει αποζημίωση για το θύμα, την οποία δικαιούται. Τελευταίο ερώτημα. Αν, για παράδειγμα, επιχειρεί μια εταιρεία σε ένα κράτος παρία ε, ποιο είναι υπεύθυνο και ποιο, δίκαιο ισχύει. Μπορεί να εφαρμοστεί, παραδείγματο χάρη, το εθνικό, το εγχώριο δίκαιο. Εγώ αναφέρθηκα στην Ιταλική νομοθεσία. Η Ιταλική νομοθεσία είναι πολύ περιοριστική για το συγκεκριμένο σημείο. Υπάρχει μια διάταξη στο ποινικό κώδικα και συγκεκριμένα ε, το άρθρο 188 το οποίο απαγορεύει την απασχόληση σε ένα ξένο κράτος. Δηλαδή στην Ιταλία αυτός ο οποίος παρέχει υπηρεσία ή εκτελεί υπηρεσία για ένα ξένο κράτος, αυτό το απαγορεύει η Ιταλική νομοθεσία και μπορεί όταν επιστρέψει από εκεί να τον συλλάβεις και να τον δικάσεις αυτόν τον άνθρωπο ή αυτή την εταιρεία. Άρα πρέπει να ισχύει το ποινικό δίκαιο. Εγώ τα λέω ξεκάθαρα τα πράγματα. Εγώ πιστεύω πιο πολύ στα εθνικά δικαστήρια και όχι στα διεθνή δικαστήρια. Σε αυτά επαφήμαι και αυτά εμπιστεύομαι για την εφαρμογή της νομοθεσίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Κυρία Μπουζάτου. Thank you. Um, I just... Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχάς θεωρώ ότι η δεσμευτική διεθνής νομοθεσία είναι το ιδανικό το οποίο και προσπαθούμε και επιδιώκουμε αλλά προσπάθησα να τονίσω στην παρουσίασή μου ότι ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό σήμερα δεν ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που καλούμαστε να ε, αντιμετωπίσουμε όπως είπε και η κυρία Λούζινγκ δεν ε, δρούμε σε ένα επίπεδο ε, ε, κράτους με συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομοθεσία για παράδειγμα Λαμβάνοντας λοιπόν αυτά υπόψη με στόχο να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τις παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων κατά το δυνατόν, αυτός ο κώδικα διοντολογίας ακριβώ αυτό που προσπαθεί να πετύχει. Για να είμαστε απόλυτα σαφεί τώρα, παρά το γεγονό ότι πρόκειται για κώδικα διοντολογίας και πρόκειται για μια διαδικασία η οποία εν μέρει υποστηρίζεται από τον κλάδο, συμμετέχουν και η κοινωνία των πολιτών και τα κράτη στη διαμόρφωσή του αναφέρεται στα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία έχουν συμφωνηθεί σε δημόσιο επίπεδο, σε δημόσιες ε, συμβάσεις ε, και στις ίδιες μας τις κοινότητες και μεταμορφώνουν αυτές τις υποχρεώσεις σε κάτι το οποίο μπορεί να ισχύσει άμεσα στις εταιρείε αυτές μέσω μιας σύμβασης. Ίσως είναι λίγο περίεργο να λέμε ότι η παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να ισούται τελικά σε μια ε, παραβίαση σημαντικού όρου. Πρέπει να γίνει έναν πρώτο τρόπο να υπάρχει μια λογοδοσία πραγματική, όπου θα, υπάρχουν, θα υπάρχει δικαστική δίωξη για παραβίαση των όρων μιας σύμβασης ως ένα πρώτο βήμα προς ε, την επίτευξη ενός δικαστικού μέσου, κάποιας λογοδοσίας. Συμφωνώ απόλυτα ότι δεν πρόκειται για την κατεξοχήν λύση. Πρόκειται για ένα βήμα ίσως, ελπίζουμε, προκειμένου τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι ανθρώπινες αξίες, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τη χρήση βίας, που πρόκειται για, πάντα, για χρήση βίας, για σκοπούς άμυνας και για την απαγόρευση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, του τράφικινγκ των ανθρωπίνων ε, ανθρώπων, απαγόρευση των χειρότερων μορφών ε, παιδικής εργασίας. Για τις εταιρείε που θα μπορούν να εφαρμόσουν ένα τέτοιο σύστημα και με την ιδέα αυτή Ελπίζουμε να αποτρέψουμε τουλάχιστον πολλές από τις παραβιάσεις αυτές προτού συμβούν. Άρα, πρόκειται για ένα ευρωδικό σύστημα για να ανταποκριθούμε σε μια ευρωδική κατάσταση όπου οι ιδιωτικοί φορείς παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες. Πρόκειται για ένα μέσο που παίρνει κάποιες δημόσιες κοινέ αξίες και τις μεταμορφώνει σε κάτι που μπορεί να εφαρμοστεί ε, ιδιωτικά και δυστυχώ θα πρέπει να αποχωρήσω πριν το τέλος της ακρόασης. Σα ευχαριστώ όμως για τις ερωτήσεις που μου θέσατε. Σα ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ. Ο καθηγητής κύριε Μπρανοβίτς. Ευχαριστώ να απαντήσω στην κυρία Λόζινγκ στα γερμανικά, αν δεν έχετε πρόβλημα. Και μάλιστα σε δύο βήματα. Το πρώτο βήμα είναι ότι θεωρώ ότι θα πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ ε, ιδιωτικών ε, επιχειρήσεων ε, στρατιωτικής ασφάλειας και αυτό που περιγράψατε. Σήμερα το πρωί που ήρθα στο Κοινοβούλιο είδα ότι υπήρχε μια ιδιωτική εσφαιρία ασφάλειας η οποία με έλεξε. Ε, δεν μπορώ να πω ότι είναι και μισθοφόρη και αυτό το λέω γιατί έχει αυτό συνέπειε για το πώς αντιμετωπίζουμε τη ρύθμιση και για το πώς ε, επηρεάζει αυτό την κρατική δομή. Καταρχάς θέλω να κάνω μια διάκριση. Είπατε και ρωτήσατε ποια είναι η βιώσιμη ε, επιρροή το, της εξωτερικής ανάθεσης ε, στην κρατική δομή. Να κάνω διάκριση μεταξύ των αποτυχημένων κρατών και των ε, αδύναμων δομών και των βιομηχανικών κρατών. Στα αδύναμα κράτη βλέπουμε συχνά ότι οι ιδιωτικές εταιρείες αναλαμβάνουν κάποιες ε, λειτουργίες οι οποίες παλιά υπήρχαν και τις είχαν αναλάβει οι σύμμαχοι. Είναι αποζημιτική ας πούμε κάπως η λειτουργία τους και είναι σαφές, είναι μάλλον απαραίτητο να ξέρουμε τι ακριβώς κάνουν. Εκπαιδεύουν, αγωνίζονται, μάχονται και μόνο με τις ερωτήσεις αυτές μπορούμε να διευκρινίσουμε ποια είναι η επιρροή στην ε, βιώσιμη οικοδόμηση κρατικών δομών και ποια προβλήματα ε, δημιουργούνται. Είναι μια εμπειρικά ανοιχτή ερώτηση. Υπάρχουν κάποιες προσεγγίσεις έρευνα, αλλά δεν έχει διευκρινιστεί το θέμα αυτό. Σε ε, κράτη ενοποιημένα τώρα έχουμε εκτελεστική εξουσία και την ανάθεση σε εξωτερικές ιδιωτικές εταιρείες έχουμε θέματα λογοδοσίας τα οποία ενδεχομένως μπορούν να συζητηθούν και στα πλαίσια ενός κώδικα διοντολογίας και υπάρχουν και θέματα απώλειας ε, ε, δυνατοτήτων μέσω διαρκούς ανάθεσης. Νομίζω ότι σε σωστά και δυνατά κράτη είναι δύο θέματα πολύ σημαντικά. Η διαφάνεια και η ολοένα αυξανόμενη διαφάνεια και είπα κινούνται προς σωστή κατεύθυνση γιατί έχουν ξεκινήσει να παρέχουν δημόσια πρόσβαση στο συνολικό όγκο των ε, συμβάσεων αυτών και το δεύτερο είναι η ρύθμιση για την λογοδοσία. Άρα η επιρροή στις κρατικές δομές εξαρτάται από το πόσο ενεργά τα κράτη αλλά και η διεθνή κοινότητα προβαίνουν σε ρύθμιση των ιδιωτικών αυτών φορέων και νομίζω ότι η ρύθμιση αυτή είναι πολύ σημαντικό θέμα, ιδιαίτερα για τα αδύναμα κράτη, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν σωστές ελεγκτικές αρχές στα κράτη αυτά. Αντιδρώντας τώρα και απαντώντας τον κύριο Γκουαλτιέρη, Μιλήσατε για έρευνες ε, κόστους προμήθειας. Κατά την προετοιμασία μου της, για την ε, ακρόαση αυτή αναζήτησα κάποια δεδομένα και άρχισα να ε, ελέγχω τις διάφορες αποστολές και και αυτό που βρήκα ήταν το τίποτα. Δεν βρήκα τίποτα. Πέρα από την αποστολή στην Παλαιστινιακή, στο Παλαιστινιακό έδαφος για το 2009 και το 2010 αν γνωρίζετε με τι γίνεται με τις ποσοτικές ερεύνες, θα ξέρετε ότι αυτά τα δεδομένα δεν επαρκούν για να γίνει μια ανάλυση ε, αποδοτικότητας κόστους. Στο επόμενο λοιπόν πράγμα που έκανα είναι ότι ζήτησα από την Διεύθυνση Προϋπολογισμών να μου στείλουν τα σχετικά δεδομένα. Έλαβα κάποια τέτοια δεδομένα, αλλά μόνο τις δαπάνες συνολικά για τις αποστολές ΚΕΠΑ. Άρα δεν έχω οποιαδήποτε ιδέα για το πόσα χρήματα ξοδεύονται σε ιδιωτική ασφάλεια, ακόμα και αν προσπάθησαν να βρω τα στοιχεία αυτά. Και αυτό ακριβώς εννοούσα, προωθώντας την ιδέα επένδυσης σε θεσμούς δημοσίων τέτοιων συμβάσεων, σε θεσμούς που θα συλλέγουν και θα κάνουν ανάλυση των δεδομένων αυτών και θα συγκρίνουν τις δημόσιες δαπάνες με την, ε, τις δαπάνες ε, ιδιωτικής ασφάλισης. Αυτό λοιπόν είναι απαραίτητο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τους συγκητές μας και ένα λεπτό διάλειμμα για να ζητήσουμε από τον κύριο Πάρκ και Κλάρκ να ανέβουν εδώ και στον κύριο Νίκολας θα ζητήσω να αναλάβει την Προεδρία. Yeah.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 We'll open the second panel. I would like to welcome the speakers for the second panel. Θα ξεκινήσω με το δεύτερο πάνελ, τη δεύτερη ομάδα ομιλητών, εκπρόσωποι των, ε, του κλάδου συγκεκριμένα. Μαζί μας είναι ο κύριος Άντι Μπέρπαρκ, ο Γενικός Διευθυντής της ε, Βρετανικής Ένωσης Ιδιωτικών Εταιριών Ασφαλείας και τον κύριο Μάικλ Κλάρκ, που είναι Διευθυντής ε, Δημόσιων Υποθέσεων G4S. Θα δώσω το λόγο στους ομιλητές για να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος. Thank Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, στην ε, σύντομη παρουσίασή μου θα ήθελα να καλύψω δύο τομείς. Ο πρώτος είναι το κατά πόσον εμείς ε, Ευρωπαίοι θα χρησιμοποιήσουμε περισσότερο τι ιδιωτικέ επιχειρήσει ασφάλεια ή επιχειρήσει σαν αυτέ τι οποίε έχουμε περιγράψει. Και δεύτερον, ποιε είναι οι τρεις προποθέσει που πρέπει να πληρούνται για αυτό το σκοπό. Να δούμε το πρώτο σημείο. Εγώ πιστεύω ότι ήδη χρησιμοποιούμε ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας και θα αυξηθεί η χρήση τέτοιων εταιριών στις, στις επιχειρήσεις μας στα προσεχή έτη. Για δύο πολύ απλούς λόγους. Κατά πρώτον, διότι υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση για τέτοιες επιχειρήσεις. Στο τέλος του ψυχρού πολέμου και τα επόμενα έτη οδήγησαν σε αύξηση διεθνικών πόλεμων, σειράξεων, συγκρούσεων και απολειών σε ανθρώπινη ζωή. Είδαμε όμως και αύξηση σε χαμηλή... Είδαμε πολύ μεγάλη ανασφάλεια και μείωση των κρατικών στρατιωτικών δυνάμεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι οι δυνατότητες ε, αντίδρασης μειώνονται ανακράτως. Άρα έχουμε μεγαλύτερη ζήτηση και μικρότερη προσφορά. Επομένως, όπως είδαμε τα τελευταία πέντε χρόνια, πιστεύω ότι και τα επόμενα 5, 10 και 15 χρόνια θα δούμε αύξηση της χρήσης ιδιωτικών εταιριών ασφάλειας αν υποθέσουμε ότι είναι σωστή η υπόθεση αυτή, εγώ πιστεύω ότι είναι, το σημαντικό ερώτημα δεν είναι αν χρησιμοποιούμε τις ιδιωτικές εταιρείε, γιατί τις χρησιμοποιούμε, η απάντηση είναι καταφατική. Το ερώτημα είναι πώς τις χρησιμοποιούμε. Από τη σκοπιά μου, τη σκοπιά των εταιριών και των γνώσεων που έχω, ως θεσμικό όργανο πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ε, εξασφαλίσει ότι πλούνται τρεις βασικοί όροι για τη χρήση αυτών των εταιριών. Πρώτος όρος, σαφήνεια των καθηκόντων. Δεύτερον, αποτελεσματική και εφαρμόσιμη ρύθμιση. Και τρίτον, είδος, ύφο των επιχειρήσεων. Ας δούμε τον καθένα όρο ξεχωριστά. Σαφή καθήκοντα. Οι ιδιωτικές εταιρείε ασφάλειας ε, σε αντιδιαστολή με τις ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες, στην αργό που χρησιμοποιούμε εμείς, παρέχουν μόνο υπηρεσίες αμυντικές, δηλαδή προστατεύουν ε, είτε ανθρώπους είτε περιουσιακά στοιχεία. Δεν επιτίθενται, δεν παρέχουν επιθετικές υπηρεσίες. Οι επιθετικές δραστηριότητες ε, παραμένουν ε, αντικείμενο των εθνικών ενόπλων δυνάμεων των κρατών. Αλλά αν δει κανεί από κοντά το όλο ζήτημα, θα καταλήξει πολύ γρήγορα στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μια γκρίζα ζώνη μεταξύ αμυντικών και επιθετικών ε, επιχειρήσεων. Και αυτοί που μελετούν ε, τι επιχειρήσει των ΗΠΑ στο Ιράκ, που ήμουν εγώ στο Αφγανιστάν, θα δουν ότι σε κάποιε περιπτώσει αυτέ οι δραστηριότητε είναι ξεκάθαρα επιθετικού χαρακτήρα. Επομένω, Ποιο είναι το βασικό καθήκον. Το πρώτο, αν εμείς Ευρωπαίοι που χρησιμοποιούμε ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας, εμείς Ευρωπαίοι λοιπόν πρέπει να ξέρουμε ξεκάθαρα για ποια καθήκοντα τις χρησιμοποιούμε και να μην τις κάνουμε να καλύψουν επιχειρήσεις οι οποίες ε, πρέπει να ε, εκτελούνται από τις ένοπλες δυνάμεις των κρατών. Δεύτερη προϋπόθεση, πολύ βασική, χρειάζεται ένα πλήρες και ξεκάθαρο ρυθμιστικό περιβάλλον και πλαίσιο. Ακούσατε τι γίνεται με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και συγκεκριμένα ακούσατε για τον Διεθνή Κώδικα Διοντολογίας που εκπώνησε η ελβετική κυβέρνηση μετά τη διαδικασία του Μοντρέ. Εγώ θα έλεγα ότι αυτός ο κώδικας διοντολογίας είναι απαραίτητο πρώτο βήμα. Δεν είναι όμως παρά αυτό και μόνο. Ένα πρώτο βήμα είναι ένα έγγραφο το οποίο φιλοδοξεί να αναφέρει πράγματα τα οποία θέλουμε να επιτευχθούν χωρίς όμως να ασχολείται το κείμενο πώς θα τα κάνουμε πράξη και ποιος θα είναι υπόλογος. Εγώ ακόμη και παρουσία ενός από τα συμβαλόμενα μέλη. Ε, πρέπει να πω ότι περισσότεροι που έχουν προσυπογράψει αυτό το έγγραφο το προσυπογράφουν χωρίς να ανησυχούν και πολύ. Γιατί αν είναι μια καλή εταιρεία, ο κύριος ε, Εξεβονίμων με σίγουρος ότι ανήκει σε μια καλή εταιρεία, ήδη ε, παρέχουν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Αν είναι όμως μια κακή εταιρεία, ξέρουν ότι δεν μπορούν να είναι υπόλογοι, άρα γιατί να μην υπογράψουν το υπογράφεις, το βάζεις και στην ιστοσελίδα το αναρτάς εκεί να το βλέπουν και τελειώνεις. Επομένως ένα πρώτο βήμα είναι αυτός ο διεθνής κώδικας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να βαθίσουμε με ταχύτερους ρυθμούς και να αναπτύξουμε, να αναπτύξουμε πρώτα σε τρεις τομείς. Πρώτος τομέας, ένα, θέλουμε ένα μηχανισμό επιβολής. Αυτός ο μηχανισμός απαιτεί την παρέμβαση των κυβερνήσεων και τη συμμετοχή των κυβερνήσεων δεν μιλάμε για καθεστώς αυτορύθμισης, γιατί κανένα από αυτά δεν είναι 100% επιτυχές στην ιστορία της Ευρώπης. Ουσιαστικά είναι ένα είδο διανοητικού άλματο αν κάποιο νομίζει ότι έτσι θα λειτουργήσει το πράγμα. Πρέπει λοιπόν οι κυβερνήσει να συμμετέχουν στην συγκρότηση αυτού του μηχανισμού επιβολή. Δεύτερον, ο Διεθνή κώδικα διοντολογία πρέπει να επεκταθεί, να διευρυνθεί και να καλύψει και τομεί που πραγματικά είναι σημαντικοί θα πρότεινα, ε, μάλλον θα έλεγα, ότι είναι λίγες οι ευρωπαϊκές χώρες που έχουν εταιρείε οι οποίες σοβαρά θέλουν να αναλάβουν παράνομες δραστηριότητες, παράδειγμα χάρη να εισβάλλουν σε μικρά αφρικανικά κράτη. Πάντως θα έλεγα ότι υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας στην Αφρική και την Ασία, οι οποίες είναι έτοιμες να προβούν σε τέτοιες δραστηριότητες. Και αν είδατε και τα στοιχεία της Σαν Μαρή, ε, στις διαφάνειες που μας έδειξε, ο κώδικας αυτή τη στιγμή ε, είναι ένας ευρωαμερικανικός κώδικας ε, ως επιτοπλίστων. Πρέπει λοιπόν να γίνει παγκόσμιος, να γίνει οικουμενικός αυτός ο κώδικας για να αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία είναι τελείως διαφορετικά στην ε, νοτίως της Σαχάρας Αφρική σε σχέση με αυτά τα οποία έχουν να αντιμετωπίσουν αμερικανικές εταιρείες ή εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου. Και ένα τρίτο μέρος της εξίωσης, αυτό που λείπει, είναι ένα είδος ελέγχου. Ο όρος ρύθμιση με ανησυχεί. Μιλάω για ένα είδος ελέγχου επί των μεμονωμένων ε, ατόμων. Υπάρχουν πολλοί παρατηρητές του κλάδου και των δραστηριοτήτων του, οι οποίοι πραγματικά εκπλήσονται ε, γιατί βλέπουν ότι ε, τελικά Υπάρχουν κάποιοι οποίοι μπαίνουν ε, για να μπουν στη λέσχη των ε, Βρυξελών, θέλουν, πρέπει να επιδείξουν ε, τα στοιχεία τους και να περάσουν από λεπτομέρεια έλεγχο, αλλά μπορώ να πάρει στο Αφγανιστάν χωρίς πρόβλημα με ένα όπλο καλάσνικο, VAK 44. Έχουμε δει διάφορα πράγματα. Αν δει κανεί τα εμπειρικά στοιχεία που ενδιαφέρουν και τους συναδέλφους, θα δούμε ότι τα περισσότερα κακά πράγματα γιατί δεν μπορώ να τα ορίσω με εμπειρικούς όρους. Τέλος πάντων, τα κακά που έχουν συμβεί τις περισσότερες φορές έχουν συμβεί ως αποτέλεσμα δράσεων μεμονωμένων ατόμων εκτός των πολιτικών ή των επιθυμιών των εταιριών τους. Επομένως, μπορεί να έχουμε μια εταιρεία που λέει όλα τα καλά πράγματα και προσπαθεί να τα κάνει και πράξη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και τα άτομα τα μεμονωμένα απαραίτητα θα εργαστούν ορθά, σωστά, άρα υπάρχει κίνδυνος να συμβούν και κάποια κακά πράγματα. Τρίτος τομέας για τον οποίο θεωρώ ότι εμείς ως Ευρωπαίοι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και στις συμβάσεις που υπογράφουμε είναι η κοινωνική συμπεριφορά. Η κοινωνική συμπεριφορά των εταιριών και των ατόμων που απασχολούνται από τις ιδιωτικές εταιρείε. Ή αν θέλετε πολιτιστική ευαισθησία, όπως θα μπορούσαμε να το πούμε. Αν εμείς θέλουμε ως Ευρωπαίοι να έχουμε παρουσία σε περιοχές όπως το Κοσφοπέδιο, η Σομαλία, η Λιβύη ίσως, ίσως τους επόμενους μήνες, τι πρέπει να κάνουμε. Εμείς έχουμε μόνο δικαίωμα να είμαστε εκεί εάν είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε το λαό των χωρών αυτών. Δεν έχουμε άλλο ηθικό δικαίωμα. Η ύπαρξή μας δεν δικαιολογείται με άλλο ε, επιχείρημα. Και αν είμαστε εκεί πρέπει να έχουμε και την ηθική υποχρέωση να εργαστούμε προς το συμφέρον του λαού Τη χώρα στην οποία θα βρισκούμε. Ε, κατά γενικό κανόνα δεν εργάζεσαι εάν... Ε, ε, ε δεν, δεν εργάζεσαι προ όφελο του πληθυσμού εάν οδηγεί ένα 4x4 και πατά ε, τα παιδιά που βρίσκονται στο διάβα σου ή τα τρομοκρατή να πεταχτούν στο πεζοδρόμιο. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι από πολιτιστικής πλευρά Σίγουρα θα χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο ιδιωτικούς ε, φορείς παροχής υπηρεσιών και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να ισχύουν αυτές οι τρεις προποθέσει που προανέφερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να σας μιλήσω για το θέμα αυτό. Να σας πω ότι είμαστε αγγλική δανέζικη εταιρεία και συμμετέχουμε στο κρηματιστήριο της Δανίας και του Λονδίνου Είμαστε ο μεγαλύτερος πάροχος ε, τέτοιων υπηρεσιών. Δραστηριοποιούμαστε σε 120 χώρες και σε 22 χώρες της κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ασφαλίζουμε και το κτίριο αυτό από τον επόμενο ε, μήνα θα ασφαλίζουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εργαζόμαστε στο αεροδρόμιο Έχουμε 600.000 ε, εργαζόμενους σε όλοι, υπαλλήλου σε όλο τον κόσμο και καταλαβαίνουμε το θέμα αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί πρόκειται για το προσωπικό μας σε περιοχές υψηλού κινδύνου με χαμηλές υποδομές όπου ο κίνδυνος και για το προσωπικό και για τον κόσμο που προστατεύουμε είναι τόσο υψηλός που ε, δίνουμε τελικά στο προσωπικό μας ε, όπλα γιατί αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη για την σωστή προστασία του κόσμου εκεί. Και φυσικά όποτε χρησιμοποιούνται όπλα χρειάζεται καλός έλεγχος και καλή νομοθεσία. Άρα αυτό αποτελεί έναν από τους τομείς που συζητούμε σήμερα για το πώς θα αριθμιστεί ο κλάδος αυτός. Πριν περάσουμε όμως τη συζήτηση αυτή να αναφέρω τι κάνει ο κλάδος ιδιωτικής ασφάλειας και τι δεν κάνει ε, και προηγούμενοι ομιλητές αναφέρθηκαν σε αυτό. Αυτό που κάνουμε είναι να παρέχουμε υπηρεσίες προστασίας. Προστατεύουμε ανθρώπους και περιουσιακά στοιχεία ανταποκρινόμενοι σε απειλές και σε... Δεν κάνουμε ποτέ επιθετικές δράσεις. Χρησιμοποιούμε ελάχιστη βία, την ελάχιστη βία σε κάθε κατάσταση μόνο τη βία που είναι απαραίτητη για προστασία των ατόμων και των περιουσιακών στοιχείων και πάντα τηρούμε το διεθνέ δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά θα έπρεπε να κάνει μια εταιρεία ιδιωτική ασφάλεια και αυτό ελπίζω ότι κάνουμε εμεί κάθε μέρα. Αυτό που δεν κάνει μια τέτοια εταιρεία είναι στρατιωτική δράση επιθετικής φύσεως. Αυτό που ανέφεραν κάποιοι και μίλησαν για μισθοφόρους. Πιστεύω ότι είναι μια τελείω διαφορετική ε, δραστηριότητα. Δεν θα πρέπει να τη συγχαίουμε με το δικό μας κλάδο. Αυτό σημαίνει ε, ότι εμπλέκεται ε, ο πάροχο αυτό σε παράνομες δραστηριότητες που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι σαφή λοιπόν ο διαχωρισμός μεταξύ του τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει να κάνει μια εταιρεία ιδιωτική ασφάλεια. Ας σκεφτούμε λοιπόν λίγο γιατί ο κόσμος χρησιμοποιεί τέτοιε εταιρείε ιδιωτική ασφάλειας. Οι βασικοί μας πελάτες είναι εμπορικές οργανώσεις, κυβερνήσεις και μη κυβερνητικοί φορείς, μη κυβερνητικέ οργανώσεις και το καθεξής. Για τους εμπορικούς οργανισμούς και για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις είναι σαφές ότι αν θέλουν να λειτουργήσουν σε δύσκολες περιοχές όπου υπάρχουν πραγματικά σωματικές απειλές είτε για την ανθρωπιστική βοήθεια, είτε για την ε, ε, εμπορική δραστηριότητα, για παράδειγμα εξόριξη, χρειάζεται κάποια προστασία και επειδή δεν έχουν τέτοια δυνατότητα, προσλαμβάνουν μια εταιρεία ιδιωτικής ασφάλειας. Το ζήτημα αυτό περιπλέκεται λίγο όταν ρωτηθούμε γιατί μια κυβέρνηση η οποία έχει ενοπλές δυνάμεις, για παράδειγμα ο ΙΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση που θεωρητικά θα είχε πρόσβαση στις ενοπλές δυνάμεις των κρατών μελών, γιατί χρησιμοποιούν λοιπόν αυτές οι οργανώσεις και οι κυβερνήσεις τέτοιες εταιρείε. Κάποιες φορές γιατί δεν έχουν κάποιες δυνατότητες, για παράδειγμα, για την αφαίρεση ναρκών, αλλά συχνά και για επιπρόσθετες δυνατότητες και ικανότητες για να απελευθερωθούν από τέτοιες ε, αρμοδιότητες, τέτοια καθήκοντα οι δικέ τους ενοπλές δυνάμεις. Για παράδειγμα, μπορεί σε μια ευρωπαϊκή αποστολή να υπάρχουν χρήματα για τα κράτη-μέλη, αλλά να μην υπάρχει ο κατάλληλος κόσμος με τις σωστές ικανότητες. Αυτά τα χρήματα μπορούν να μετατραπούν ε, μέσω ανάθεση σε μια ιδιωτική εταιρεία σε υπηρεσίες ασφαλείας. Και γενικά είμαστε πιο αποτελεσματικοί από πλευράς κόστους, από τις ενοπλέ δυνάμεις, τις κρατικές, γιατί παρέχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο, μια πολύ συγκεκριμένη υπηρεσία και το προσωπικό μας είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για τις υπηρεσίες αυτές. Αντίθετα με τις ενοπλέ δυνάμεις ενός κράτους που έχουν μια τεράστια βάση και ένα τεράστιο εύρος στην εκπαίδευσή τους, άρα το κόστος τους τίνει να είναι πιο υψηλό όπως είπε και ο Άντι προηγουμένως, με τις περικοπές ε, στον προϋπολογισμό για την άμυνα, πολύ απλά δεν υπάρχουν ενοπλές δυνάμεις για την προστασία που θα χρειαζόταν. Παίρνοντας λοιπόν τώρα στο θέμα της ρύθμισης των κανονισμών, καταλαβαίνουμε ότι ο κλάδος πρέπει να ρυθμιστεί καταλήλως. Κάποιες χώρες το πράττουν αυτό, οι ε, όλο και πιο πολύ το κάνουν θέτοντας αυστηρούς όρους στις συμβάσεις το Ηνωμένο Βασίλειο προ αυτήν την κατεύθυνση κινείται και αυτό. Αλλά υπάρχουν μεγάλα χάσματα σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση και νομίζω ότι όλοι το αναγνωρίζουμε αυτό. Μιλήσαμε για κάποια ενδεχόμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Υπάρχει ένα θέμα για το κατά πόσο θα ήταν αποτελεσματική η νομοθεσία αυτή για τον κλάδο αυτό, γιατί όπω συζητήσαμε, οι πιο πολλέ εταιρείε στον κλάδο αυτό δραστηριοποιούνται εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο πολλέ εταιρείε έχουν και έντρα εκτό Ένωση. Νομίζω ότι από τις εταιρείες που έχουν προσυπογράψει τον Διεθνή Κώδικα, το 43% μόνο έχει έδρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα ένα μεγάλο κομμάτι είναι εκτός. Και ουσιαστικά όλες τους οι δράσεις θα είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα είτε υπάρχει Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, δεν ξέρω αν θα ήταν αποτελεσματική. Όπως είπε και ο κ. Μπασάτου, η κυρία Μπαζάτου, προσπαθήσαμε να γεμίσουμε, να πληρώσουμε αυτό το χάσμα με έναν διεθνή κώδικα, ο οποίος νομίζω περνάει πέρα από τα όρια της αυτορύθμισης και συμπεριλαμβάνει και τις κυβερνήσεις, ελεύθερε κυβερνήσεις ε, κατά κανόνα, τι οργανώσει της κοινωνία των πολιτών, Human Rights Watch και άλλες οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα συμμετέχουν στην κατάρτιση του κώδικα αυτού και εγώ συμμετέχω στην ε, Επιτροπή για την εφαρμογή ενός μηχανισμού ε, εφαρμογής. Γιατί όπως είπε ο, κώδικ, ο Άντι, αυτός ο κώδικας στην παρούσα φάση είναι μια φιλοδοξία για το πώς θα έπρεπε να, να συμπεριφέρεται ο κλάδος. Δεν υπάρχουν ακόμα κυρώσεις, αλλά... Όλοι θεωρούν ότι θα έπρεπε να υπάρχουν κυρώσεις, θα πρέπει να υπάρχει σαφήνεια για το αν μια εταιρεία συμμορφώνονται ή όχι με τον κώδικα και αν δεν συμμορφώνονται να υπάρχουν κυρώσεις και να δημοσιοποιείται το γεγονός αυτό, να υπάρχει ένας μηχανισμός μέσω του οποίου θα μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις και ο κώδικας, ξέρετε, είναι πάρα πολύ ευρύς. Περιλαμβάνει την επιλογή, κατάρτιση του προσωπικού, τη διαχείριση του προσωπικού, τη χρήση βίας, τη χρήση όπλων, το γενικό σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την αναφορά ε, περιστατικών και πολλά άλλα τέτοια ζητήματα τα οποία αν εφαρμοστούν θα ε, έχουν μια φορά σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες ε, των εταιριών επιτόπου. Ένα τελευταίο στιγμή τώρα για κάποια θαλάσσια ζητήματα τα οποία ανέφεραν και κάποια από τα μέλη της Επιτροπής. Καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ένα τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται όλο και πιο πολλοί οι ιδιωτικές εταιρείες δεδομένων και των προβλημάτων με την πειρατεία, ιδιαίτερα στι ακτέ τη Σομαλία. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ περίπλοκο το θέμα αυτό από πλευρά νομικών συστημάτων. Ποιο νομικό σύστημα ισχύει, ποια είναι η κατάλληλη χρήση βία και ούτω καθεξή. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ανάγκη για ρύθμιση. Ο κώδικα δεν τα αποκρίνεται στι ανάγκε αυτέ, αλλά πρόκειται για το επόμενο θέμα στον κατάλογο των ε, στοιχείων που θα πρέπει να διαπραγματευτούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Λίγο ο Πρόεδρος. Κάποιες ερωτήσεις να ακούσουμε, κάποιες παρατηρήσεις ίσως. Η κυρία Μπράβνερ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τους δύο για τις παρουσιάσεις σας. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Ένα γενικό σχόλιο. Είπατε ότι γιατί να μας βοηθήσει η ευρωπαϊκή νομοθεσία όταν ε, μιλάμε μόνο για ένα 43%. Νομίζω ότι είναι σημαντικό τμήμα αυτό το 43%. Σχεδόν το ίμιση θα ρύθμιζα. Θα ρύθμιζε η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτή είναι όμως ε, η εντύπωση που έχουμε ε, και για πολλά άλλα θέματα. Για παράδειγμα, για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή. Αν ρωτιόμαστε γιατί να ξεκινήσουμε εμεί ω Ευρωπαίοι, γιατί μα ακολουθούν οι υπόλοιποι. Αν μπορούμε κάτι να κάνουμε, καλύτερο είναι από το να μην κάνουμε τίποτα. Μία ερώτηση έχω να κάνω και το θέμα της λογοδοσίας και αυτό το χάσμα που αναφέρεται ότι υπάρχει για τα άτομα. Γιατί είπατε ότι ακόμα και αν οι εταιρείε δεσμευτούν κάποια άτομα, κάποιοι υπάλληλοι στο ιστορικό των εταιρεών μπορεί να μην συμμορφωθούν. Άρα, ποιο είναι ο πιο αποτελεσματικό τρόπος να υπάρχει λογοδοσία για τις ενέργειες του καθενό κοιτώντας τα μεμονωμένα άτομα, θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει πριν διαπράξουν ε, μία πράξη και τι συμβαίνει μετά. Αν για παράδειγμα χρησιμοποιήσουν αλκοόλ και πάρουν ναρκωτικά και σκοτώσουν κάποιον, έχουν διαπράξει ένα έγκλημα υπάρχουν θέματα, γιατί αν διαπράξουν ένα τέτοιο έγκλημα στο Αφγανιστάν ή στο Ιράκ σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, μπορεί να μην υπάρχει σύστημα να τους δικάσουν. Αλλά πολλές χώρες, και συγχωρέστε μας γιατί δεν είμαι δικηγόρος, αλλά έχουμε μαζί ένας ε, καθηγητή, υπάρχουν ε, κάποιες τέτοιες διατάξεις εκτός ε, ε, περιφέρειας. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό για το Ηνωμένο Βασίλειο, αν ένα Βρετανός διαπράξει έγκλημα, μπορεί να διωχθεί σε βρετανικά δικαστήρια. Νομίζω για τους Γερμανούς ε, αυτό περιλαμβάνει οποιοδήποτε ε, έγκλημα. Για οποιοδήποτε έγκλημα μπορεί ένας Γερμανός επίκος να διωχθεί στη Γερμανία αλλά νομίζω ότι αυτό που απασχολεί τους πιο πολλούς είναι για τα πρότυπα ε, πρόσληψης για το πώς επιλέγονται αυτοί οι άνθρωποι και κατά πόσον υπάρχει κάποιος καλύτερος τρόπος προκειμένου να μην ε, ε, προσληφθεί κάποιος ο οποίος ενδεχομένω να παρουσιάζει προβλήματα και οι εταιρείε ασφαλώς είναι 100% υπέρ ενός τέτοιου συστήματος δεν θέλουν να προσλαμβάνουν άτομα που θα παρουσιάσουν προβλήματα πώς θα εφαρμόσουμε όμως ένα τέτοιο σύστημα και το μεγαλύτερο η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων ε, ελέγχου σε περιπτώσεις ε, διαταραχών άγχους, γιατί σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις που μιλάμε για τέτοια άτομα, μιλάμε για πρώην στρατιωτικούς, οι οποίοι έχουν εκτεθεί σε διάφορα περιστατικά στην στρατιωτική τους καριέρα. Το ερώτημα λοιπόν που ανακύπτει είναι κατά πόσο ο έλεγχος των ιδιωτικών εταιριών μπορεί να βελτιωθεί με τέτοιο τρόπο, και σε τέτοιο βαθμό προκειμένου να καταστεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τις ίδιες τις εταιρείες. Όποιος έχει κοιτάσει τέτοια θέματα θα αποδεχτεί ότι φυσικά ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε τέλειοι στο σύστημα αυτό, αλλά όπως είπατε το γεγονός ότι η Ευρώπη Είπατε ότι η Ευρώπη μπορεί να κάνει κάτι από το να μην κάνει τίποτα. Ε, το ίδιο ισχύει και εδώ. Αν μπορούμε ε, να αποφύγουμε να προσλάβουμε κάποια άτομα τα οποία έχουν πρόβλημα με το σύστημα αυτό, ε, δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να προσπαθήσουμε. Να προσθέσω και εγώ κάτι ό,τι προσπαθούμε να κάνουμε εδώ ή με το Διεθνή Κώδικα Δεοντολογίας δεν μπορεί να υποκαταστήσει σε καμία περίπτωση το εθνικό δίκαιο που διέπει τις περιφορές των ανθρώπων. Αν μιλάμε για ένα διαλυμένο κράτος, ένα κράτος παρία, εκεί πάντοτε θα υπάρχει πρόβλημα επιβολής της νομοθεσίας. Λίγα πράγματα μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά που είπατε είναι επίκαιρα, σοβαρά, αλλά υπάρχουν θεμελιώδη προβλήματα τα οποία δεν μπορούμε να λύσουμε εμείς ε, από τον κλάδο μας. Υπάρχει κάποιος άλλος που δεν θέλει το λόγο. Κύριε Μπραντ. Ναι, θα ήθελα να επεκταθείτε λίγο, αν μπορείτε, σε σχέση με αυτή τη Βρετανική πρωτοβουλία, την νομοθετική που αναφέρατε. Απάντηση. Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε πρόσφατα ότι μίλησαν για αυτορύθμιση, αλλά νομίζω ότι υπερβαίνει την αυτορύθμιση. Δηλαδή, μιλάμε για μια συνεργασία με τον κλάδο του Ηνωμένου Βασιλείου για την παρακολούθηση ενό κώδικα διοντολογία που θα αντικατοπτρίζει εκ του σύνεγγυ τον διεθνή. Δηλαδή, μιλάμε για συμμόρφωση με τον κώδικα που θα εντάσσεται στη συμβάση, στα συμβόλαια των εταιριών και δύο των μεγάλων ιδιωτικών εταιριών ασφαλή που χρησιμοποιεί η Βρετανική κυβέρνηση. Δεν θα είναι δηλαδή κάτι καινούριο, θα είναι κάτι μεταξύ αυτορύθμιση και νέα νομοθεσία. Νομίζω ότι αναγνωρίζουν ότι η νομοθεσία ε, σε μια εθνικό επίπεδο ε, δεν είναι ε, κάτι εύκολο, γιατί πολλές εταιρείες μετακινούνται από τη μια χώρα στην άλλη. Αν μια χώρα γίνει ιδιαίτερα δυσχερής ως προς το να εκτελούν εκεί τη δραστηριότητά τους, θα μετακατασταθούν σε κάποια άλλη χώρα και σε μια διαφορετική δικαιοδοσία, όπου δεν θα διέπονται από το δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου, για παράδειγμα. Δηλαδή οι χώρες της Ένωσης είναι εύκολες. Όχι απαραίτητα εντός Ένωσης είναι απάντηση. Καθά εκεί είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θέλουν τον λόγο. Θέλω να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους μας για τις πληροφορίες που μας έδωσαν σήμερα. Ελπίζουμε να σας ξαναδούμε σύντομα στην Επιτροπή μας στο πλαίσιο μιας νέας ομάδας ομιλητών και θα διακόψουμε τώρα μέχρι να έρθει στο βήμα το τρίτο πάντελ. Θα περάσουμε στο τρίτο πάνελ ομιλητών, όπου θα ακούσουμε τη θεσμική άποψη. Οι μιλητέ μα είναι από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Μαζί μα είναι ο κύριο Κι Κλόμπεν-Χάουερ, διοικητή ε, αστικών επιχειρη... πολιτικών μάλλον επιχειρήσεων και ο κύριος Πάτρικ Τσάιλτ ε, που είναι ευθύνων σύμβουλος για την ε, διοίκηση και τα οικονομικά. Να δώσω μέσω στο λόγο στους προσκεκλημένους μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε και πάλι μεγάλη μου τιμή να σας ε, μιλώ. Um, για δεύτερη φορά σήμερα για το θέμα εταιριών ιδιωτική ασφάλεια και από ό,τι κατάλαβα ήταν ήδη γεμάτη η μέρα σα το απόγευμά σα με συζητήσει σχετικέ Για μα το θέμα δεν είναι καθόλου απλό. Να σα δώσω κάπω τις αδρέ γραμμέ. όμως. Καταρχά, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να ιδρύσει αποστολές ε, και πά σε τομείς όπου υπάρχει θέμα ασφάλειας, όπως το Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Αυτή είναι μια πρώτη πραγματικότητα και από την πραγματικότητα αυτή προκύπτει ότι η πρώτη προτεραιότητά μας θα πρέπει να είναι να διασφαλίσουμε, ε, να φροντίζουμε το προσωπικό το οποίο έχουμε αναπτύξει στις περιοχές αυτές. Πέρα από τα ηθικά ζητήματα, υπάρχουν και νομικές συνέπειες σε περίπτωση αποτυχίας σε, σε ό,τι αφορά την φροντίδα αυτή και την αποτελεσματική προστασία των ατόμων τα οποία αποστέλουμε σε μια τέτοια αποστολή. Η πραγματικότητα είναι η εξής. Υπάρχει πολύ περιορισμένος αριθμός δυνατοτήτων για την προστασία των ατόμων αυτών. Καταρχάς, ένα κράτος μέλος θα μπορούσε να φροντίσει το θέμα αυτό. Κατά δεύτερον, η ίδια η αποστολή θα μπορούσε να αναθέσει ένα προσωπικό ασφαλείας στο ιστορικό της αποστολής. Τρίτη λύση θα ήταν να προσληφθεί μια εταιρεία ιδιωτικής ασφάλειας και τέταρτη δυνατότητα, σε περίπτωση που δεν λειτουργούσαν οι υπόλοιποι, είναι να κλείσει η αποστολή. οι εγχώριες ε, αστυνομικέ δυνάμεις ε, φαίνεται ότι δεν μπορούν να εγγυηθούν αποτελεσματικά την ασφάλεια. Και μακροπρόθεσμα αυτό μπορεί και να αλλάξει, αλλά ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε στην εκάστοτε αποστολή είναι γιατί συνήθως βρισκόμαστε σε ένα κράτος παρεία. Άρα, βρισκόμαστε εκεί ακριβώς επειδή οι αστυνομικέ δυνάμεις δεν είναι σε θέση να αντιδράσουν. Άρα δεν μπορούμε να στηριχτούμε στις αστυνομικέ δυνάμεις αυτές για να μας παρέχουν ασφάλεια αναγνωρίζουμε ότι από νομική, πολιτική άποψη υπάρχουν προκλήσεις και συμφωνούμε με αυτά που αναφέρατε και οι μελέτες κόστους ωφέλους στην περίπτωση του Αφγανιστάν καταδεικνύουν ότι ίσως οι εταιρείε εθνικής ασφάλειας είναι η πιο φθηνή λύση στην προκειμένη περίπτωση. Υπάρχει και φυσικά και το θέμα της αφικτότητας, γιατί οι υπόλοιπε λύσεις δεν είναι απαραίτητα εφικτές. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική αρχή. Το περιεχόμενο της αποστολής καθορίζει τα, τις δαπάνες ασφάλειας. Και όταν λέω το ε, όλο, ε, εννοώ μάλλον την εντολή της αποστολής, και φυσικά το περιβάλλον ασφαλείας αποτελεί ένα επιπλέον, ένα επιπλέον στοιχείο, το οποίο πολλές φορές είναι υψηλού κινδύνου και εχθρικό. Άρα αυτά καθορίζουν το τι θα πρέπει να κάνει η αποστολή και πώς θα πρέπει να κινηθεί ο κόσμος, το προσωπικό και καθορίζουν φυσικά και τις δαπάνες και την κατάσταση προς την ασφάλεια. Αναγνωρίζουμε ότι ίσως να υπάρχουν ε, αμφιβολίες για την ε, το, την προέλευση των εταιριών προσπαθούμε συνολικά να ελαχιστοποιήσουμε αυτές τις ανησυχίες μέσω διαφανών διαδικασιών ε, ανάθεσης συμβάσεων, μέσω καλής διαχείρισης των συμβάσεων και με, με ε, απαιτώντας δέουσα επιμέλεια από τους συμβαλόμενους. Τέλος, η εξωτερική υπηρεσία, η υπηρεσία εξωτερικής δράσης, τολμώ να πω, ότι ακολουθεί μια ενιαία προσέγγιση για την προστασία του προσωπικού σε αποστολέ. Ωστόσο, επειδή είναι διαφορετικό το συγκείμενο κάθε αποστολή συνεπάγεται και διαφορετικό κόστος. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να κλείσω την πρώτη μου γενική παρέμβαση και να δώσω τον λόγο στον συναδελφό μου. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Κέις. Να προσθέσω κι εγώ μια προοπτική από πλευράς της των αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι και αποστολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου αντιμετωπίζουμε πολύ παρόμοιες προκλήσεις σε ό,τι αφορά την παροχή της κατάλληλης ε, ασφάλειας για το προσωπικό μας, τα κτηριά μας και για τα άλλα περιουσιακά μας στοιχεία σε άλλες χώρες για αποστολές και πα. Και ακολουθούμε ευρέως παρόμοιες προσεγγίσεις για την αξιολόγηση κινδύνων και την αξιολόγηση των ε, αναγκών ως προς την ασφάλεια του προσωπικού μας. οι χώροι όπου συνεργαζόμαστε με ιδιωτικές εταιρείες είναι όπου υπάρχει ο πλέον υψηλός κίνδυνος, όπου υπάρχουν υπηρεσίες για την προστασία του προσωπικού των οικειών τους και σε κάποιες περιπτώσεις προστασία του επικεφαλής της αποστολής. Πρόκειται για συμβάσεις τις οποίες συνάπτουμε με τις εταιρείε ασφάλειας μετά από διαδικασίες ε, ε, ανάθεσης ε, που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία δημοσιοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως και για τις αποστολές ΚΕΠΑ οι συμβάσεις αυτές και φυσικά εξαρτούνται πάντα από τις συγκεκριμένες ανάγκες στην κάθε χώρα και λαμβάνουμε υπόψη και τις δραστηριότητες της αποστολής. Η υπηρεσία εξωτερική δράση ασφαλώ αποτελεί μια καινούργια οργάνωση. Νομίζω ότι είναι εξαιρετική λοιπόν η στιγμή για την διοργάνωση τη ε, ακρόαση αυτή, προκειμένου να εξεταστούν οι διάφορε λύσει που έχουμε στη διάθεσή μα. Σε μια χρονική στιγμή που και εμεί οι ίδιοι εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο στο μέλλον θα φροντίσουμε για να καλυφθούν οι ανάγκες ασφάλειας του προσωπικού μας. Είτε μιλάμε για προσωπικό σε αποστολές, είτε μιλάμε για προσωπικό στα πλαίσια αποστολών και ΕΠΑ. Όπως σας είπα, είναι παρόμοια διαδικασία που ακολουθείτε, αλλά πρόκειται για κάτι το οποίο δεδομένη της έμφασης που έχει θέσει κάθε άστον στην διασφάλιση της ασφάλειας για το προσωπικό μας σε πολύ συχνά, όπως είπα, δύσκολες καταστάσεις. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο θα πρέπει να ολοκληρώσουμε επιτυχώς και είμαι βέβαιος όπως θα προχωράμε στην ανάπτυξη της νέας ε, υπηρεσίας, ε, το τμήμα υπηρεσία ασφάλειας της υπηρεσίας θα διασφαλίσει τη βέλτιστη ασφάλεια του προσωπικού και των περισσιακών στοιχείων και φυσικά θα επιλέξουμε τη λύση που θα κοστίσει λιγότερα στον κοινωνικό προϋπολογισμό. Ευχαριστώ. Any questions or ερωτήσεις, παρατηρήσεις. Παρακαλώ. Θέλω να σας ξανακαλωσορίσω, γιατί σας είδαμε και το πρωί. Σας ευχαριστώ πάντως που είστε εδώ. Έχω λίγες ερωτήσεις, γιατί είπατε ότι η πρώτη επιλογή είναι την προστασία να το αναλάβουν τα κράτη-μέλη. Πόσο συχνά τελικά ε, το καταφέρνετε αυτό, έτσι για να καταλάβουμε λίγο πόσο πρόθυμα τα κρατημέρια και πόσο συχνά του ζητάτε να λάβουν την προστασία. Δεύτερο ερώτημα. Όταν ε, τέλος πάντων ε, έχετε συμβόλαια με ιδιωτική εταιρεία, τι σύστημα υπάρχει, πώς αξιολογείτε τους ε, προμηθευτές. Και το τρίτο ερώτημα. Έχετε έναν ενοποιημένο διαγωνισμό, μια πρόσκληση υποβολής προσφορών ή έχετε συμφωνίες ε, πλαίσιο με κάποιες εταιρείες που έχουν ένα καλό ιστορικό ή επιλέγετε το φθηνότερο προμηθευτή. Ποια διαδικασία ακολουθείτε και με βάση ποιο κώδικα διοντολογία δραστηριοποιούνται αυτέ οι εταιρείε. Επιλέγεται παραδείγματο χάρη εταιρείε ε, που έχουν ε, υπογράψει το διεθνή κώδικα διοντολογία και μόνο αυτέ τι εταιρείε επιλέγεται ή υπάρχουν άλλα κριτήρια για την επιλογή τη ιδιωτική εταιρεία ασφάλεια. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις που μου κάνατε. Σε ό,τι αφορά τα κράτη-μέλη. Ποιο είναι το θέμα. το απαιτούμενο προσωπικό είναι πάρα πολύ ισχνό. Τα είδη τώρα των καθηκόντων που θα πρέπει να εκτελεστούν φύλαξη, προστασία είναι καθήκοντα που δεν ενδιαφέρονται να ασκήσουν τα ίδια τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη ενδιαφέρονται να στέλνουν στις αποστολές πιο υψηλό βαθμό προσωπικό αν θέλετε για να κάνουν τη διαφορά. Άρα κατά κανόνα τους πιο χαμηλόβαθμους ε, αξιωματούχους τους δεν τους στέλνουν σε αποστολές. Δεν τους ενδιαφέρει. Επομένως, εκεί έχουμε ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι ότι, ναι, βέβαια, επειδή και ο εξοπλισμός και η διάθεση των απαραίτητων προσώπων και ό,τι απαιτείται τέλος πάντων συνεπάγεται υψηλό κόστος για τα κράτη-μέλη και επειδή ο προεπολογισμός ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα αυτό, για τις αποστολές και ουσιαστικά επιδοτεί ένα μέρος μόνο, χρηματοδοτεί ένα μέρος, ασκούμε εμείς αυτή την πολιτική. διότι ξέρουμε πώς έχει κατάσταση, ξέρουμε ότι υπάρχει απροθυμία από πλευράς κρατών μελών να αναλάβουν αυτά τα καθήκοντα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το σύστημα προσλήψεων, δεν είμαι και πολύ πέρα αυτού του συστήματος, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει επιλογή εταιριών με βάση τις φήμες τους, αν θέλετε, και υπάρχει ένα συμβόλαιο στο οποίο γίνεται αναφορά σε ζητήματα όπως ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο σε ένα συμβόλαιο να αναφερθεί κανείς ρητά ε, στο Διεθνικό Δικαδεοντολογίας επειδή δεν είμαστε βαλωμένο μέλο, αλλά μπορούμε να μιλήσουμε για τη δέουσα επιμέλεια, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κάπω έτσι παρακάμπτουμε αυτό το πρόβλημα και έτσι αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Και βέβαια, οι εταιρείε πρέπει να έχουν εύρωστη χρηματοοικονομική κατάσταση πρέπει να έχουν ε, ένα διοικητικό συμβουλίο που να απαρτίζεται από εξέχοντα άτομα, να είναι ασφαλισμένα, να μπορούν να καλύψουν, ε, έχουν ευθύνη δηλαδή κάλυψη σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά. Όλα ό,τι συνιστούν μια καλή εταιρική διακυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά αυτές τις ενοποιημένες, τους ενοποιημένους διαγωνισμούς που είπατε, στην ΚΕΠΑ, η αποστολή είναι αυτή η οποία κάνει το συμβόλαιο. Επομένως, υπ' αυτήν την έννοια δεν υπάρχει ένα σύστημα ενοποίησης όλων των συμβολέων για όλες τις αποστολές. Για να, απαντήσουν, ίσως θα, για να απαντήσω θα έπρεπε πρώτα απ' όλα να συμβουλευτώ εμπειρογνώμονες, αλλά κάτι μου ψιθυρίζουν από δίπλα. Α, ναι, ακριβώ, ακριβώ. Υπάρχουν συμβάσει, συμβόλαια πλαίσιο για θέματα που έχουν να κάνουν με εξοπλισμού, παραδείγματο χάρη τεθωρακισμένα, αλλά όχι για τι ιδιωτικέ εταιρείε ασφάλεια. Και αυτό μεταξύ άλλων, γιατί υποθέτω ότι η κατάσταση τη ασφάλεια διαφέρει άρα πολύ από τη μία περιοχή στην άλλη. Η κατάσταση στην Καμπούλ δεν είναι το ίδιο με τη Βαγδάτη. Είναι δηλαδή ουσιαστικά προσαρμόζεται, εξατομικεύεται ανάλογα με το θέτρο επιχειρήσεων. Παραδείγματο χάρη στην Βαγδάτη, στη, η Βρετανική πρεσβεία παρέχει ένα μεγάλο μέρος της ασφάλειας της αποστολής. Άρα για την κινητή ασφάλεια κυρίως εμείς συμπληρωματικά παρεμβαίνουμε. Έχουμε συμβόλαια με τα κράτη-μέλη τα οποία είναι εκεί και μπορούν να μας παράσχουν και φιλοξενία στην πράσινη ζώνη. Άρα είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση από την ε, μία χώρα στην άλλη και από την μία περιοχή στην άλλη. Αυτή είναι η απάντηση που έχω να σας δώσω. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι. Uh, Θα μπορούσα ίσως και εγώ να προσθέσω κάτι σε ό,τι αφορά τις αντιπροσωπείες. Την ίδια εμπειρία έχουμε και εμείς σε σχέση με το επίπεδο ενθουσιασμού και ετοιμότητας που βλέπουμε από τα κράτη-μέλη ε, για να παράσχουν αυτά ε, τις υπηρεσίες αυτές από τους εθνικούς πόρους που διαθέτουν. Παραδείγματο χάρη στην αποστολή ε, και ΚΕΠΑ στη Βαγδάτη και στο Ιράκ επίσης έχουμε μια τέτοια περίπτωση. Επειδή μοιραζόμαστε τα γραφεία μας με την Βρετανική Πρεσβεία, εποφελούμεθα της ε, όλης οργάνωσης ασφάλειας της πρεσβείας. Και αυτό είναι πολύ... Ε, και είναι και ένα θέμα κόστους. Δηλαδή αναλαμβάνει κόστος και η Βρετανική Πρεσβεία. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την ε, περιπτώσεις αυτές με περιπτώσεις που εμείς αναλαμβάνουμε την ασφάλεια και φυσικά κάνουμε και την ε, δέουσα αξιολόγηση των συμβολέων και αντλούμε τα διδάγματα από τις αξιολογήσεις αυτές. Οπότε, εν συνεχεία, εκπονούμε και ε, τη συγγραφή υποχρεώσεων για, τις προσεχείς, ε, για τους προσεχείς διαγωνισμούς μας. Έχουμε αρκετή εμπειρία και πραγματικά έχουν βελτιωθεί σημαντικά οι συγγραφές υποχρεώσεων πάντα με βάση την προηγούμενη εμπειρία που έχουμε αποκομίσει. Ουσιαστικά αυτό το οποίο θέλουμε είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι εταιρείε είναι και από τεχνική πλευρά επαρκώ ικανέ για να παράσχουν τι υπηρεσίε που ζητούμε, αλλά και από την άλλη πλευρά διαθέτουν συστήματα δημοσιονομική διαχείριση και διακυβέρνηση ε, που ε, αντιστοιχούν στα ανώτατα δυνατά πρότυπα. Αυτό το οποίο θέλω να σχολιάσω είναι ότι ο ρόλος, τα καθήκοντα της ιδιωτικής εταιρείας ασφάλειας είναι να παρέχει παθητική ασφάλεια, την προστασία δηλαδή των προσώπων και των κτηρίων μας και να μην έχει άλλο ενεργό ρόλο. Από πλευράς πολιτικής σε ό,τι αφορά ομαδικές, ε, ομαδικούς διαγωνισμούς, ε, group tenders. Αυτή τη στιγμή έχουμε δρομολογήσει έναν ε, μεγάλο διαγωνισμό με διάφορες παρτίδες που θα έχει ως αποτέλεσμα τη σύναψη μιας σύμβασης πλαισίου, θα τον λέμε παγκόσμιο διαγωνισμό, όπου θα έχουμε μια δέσμη συμβάσεων που συνάπτουμε σε διάφορες περιοχές, σε διάφορα μέρη. Και αυτό το προτιμούμε παρά την προσέγγιση κατά περίπτωση που ακολουθήσαμε κατά το παρελθόν. Αυτή είναι μια εξέλιξη λοιπόν, είναι κάτι καινούριο για μας μια νέα εμπειρία. Βέβαια, οι καταστάσεις και οι ανάγκες ανάλογα με την περιοχή διαφέρουν. Αυτό είναι σαφές. Όπως είπε και ο Κις, απουσία αριθμιστικού πλαισίου, αυτό που φροντίζουμε εμείς είναι η τήρηση των αρχών μας από τις ε, εταιρείε και γι' αυτό συμπεριλαμβάνουμε αυτούς τους όρους και αυτές τις προϋποθέσεις ε, στις συμβάσεις μας. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις? Όχι. Και πάλι κυρία Μπραντ, Συγγνώμη που επανέρχομαι. Είστε Βρετανός κύριε Τσάιλτ. Ε, με τρέλανε που σας ήρθε πρώτα η γαλλική λέξη για τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα ήθελα να επανέλθω σε κάποια από αυτά που αναφέρατε. Μιλήσατε για αυτή τη συμφωνία πλαίσιο. Που είπατε ότι δεν αντιτίθεται στην ιδέα, ε, μάλλον δεν αντιτίθεται στο ότι υπάρχουν διαφορετικές καταστάσεις επιτόπου και έχουμε και πάρα πολλά σενάρια τα οποία πρέπει να επεξεργαστούμε. Επομένως δεν ξέρω κατά πόσον τελικά οι εταιρείε ε, έχουν να παρέχουν τελείω διαφορετικά υπηρεσίε ανάλογα με την περίπτωση. Χαίρομαι που προχωράτε εσεί προ μια πιο ομαδοποιημένη προσέγγιση. Βέβαια, ε, σε ό,τι αφορά την εξωτερική ανάθεση, τελικά τα κράτη-μέλη πληρώνουν, όπως και να έχει. Γιατί και ο κοινοτικός προβληματισμός από αυτούς προέρχεται. Άλλοι πληρώνουν περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Αλλά ίσως θα πρέπει να δούμε ε, εκ νέου τον όλο αυτό μηχανισμό χρηματοδότησης για να είναι ισοβαρής. Και να δούμε και αν είναι πιο ε, οικονομικό, αποδοτικό να χρησιμοποιούνται υπηρεσίες των κρατών μελών. Είπατε κάτι για το Ιράκ. Είπατε ότι χρησιμοποιείτε κάποιες βρετανικές ε, εγκαταστάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι πληρώνει πολύ μεγαλύτερο τίμημα από τους δανούς σε σχέση με το κτίριο το ίδιο. Γιατί γίνεται αυτό, πώς το δεχόμαστε και ποιο, ποια είναι η σχέση κόστους ε, αποδοτικότητας, κόστους αποτελεσματικότητας. Μου με εκπλήσει που διαφορετικά, ε, διαφορετική είναι η τιμή που πληρώνει το Ηνωμένο Βασίλειο, διαφορετική Δανία και διαφορετική Ευρωπαϊκή Ένωση για το ίδιο κτίριο. Δεν είναι αποδεκτό αυτό. Και ένα άλλο ερώτημα σε ό,τι αφορά τον ε, κώδικα διοντολογίας. Από ό,τι κατάλαβα είναι ένας ε, κώδικας διοντολογίας που υπογράφεται από εταιρείε, άρα όχι από το κράτο, όχι από το Ηνωμένο Βασίλειο. Άρα δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εσεί ω κριτήριο αυτόν τον κώδικα. Είπατε ότι δεν είσαι συμβαλόμενο μέρο. Αλλά αυτό μπορούμε να το αποκλείσουμε ότι μπορεί να γίνει. Παραμένει το ερώτημά μου πώς αυτός ο κώδικας διοντολογίας χρησιμοποιείται από εσάς στο πλαίσιο πρόσκλησης ε, υποβολής προσφορών. Και σε σχέση με την αξιολόγηση των προσφορών είπατε ότι επανασυγγράφεται τη συγγραφή υποχρεώσεων και είναι ευχάριστο που το ακούω αυτό. Αλλά άλλο ρωτάω, πώ αξιολογείτε τι εταιρείε. Σε σχέση δηλαδή με το ποια εταιρεία θα χρησιμοποιήσετε την επόμενη φορά. Έχετε μία κόκκινη λίστα ε, απαγορευμένων εταιρείων, δηλαδή που δεν θα ξαναχρησιμοποιήσετε. Δηλαδή έχετε κάποιες εταιρείε ε, στη μαύρη λίστα, θα το έλεγα καλύτερα, που δεν θα τις ξαναχρησιμοποιούσατε. Δεν λέω για τη συγγραφή υποχρεώσεων πώ την ε, συντάσσει την επόμενη φορά, αλλά τι εταιρείε επιλέγει. Και σε ό,τι αφορά το προσωπικό. Το προσωπικό αγοράς. Πώς το εκπαιδεύεται σε σχέση με όλα αυτά τα ζητήματα και σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, το κενό λογοδοσίας, ευθύνης, ε, εκπαιδεύονται συγκεκριμένα, ξέρουν τι είναι ο κώδικας δεντολογίας. εκπαιδεύονται, αυτό είναι το ερώτημά μου ουσιαστικά. Και τέλος, υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο αξιολόγησης κινδύνων που έχει η υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Ένα γενικό, λέω, ένα χώρο. Sorry, a lot of questions, but I think... Yeah. Ναι. Right. Πολλές ερωτήσεις. Besides, you can answer. Thanks. Αλλά θα μπορούσατε να απαντήσετε. If I can take them yeah, in reverse order and, and help me out when it becomes difficult. <laughs> Mike, is it working? thank you. I'll take reverse order. Yes, there is. Αντίστροφα θα απαντήσω στις ερωτήσεις. Ναι, υπάρχει ένα πλαίσιο αξιολόγηση κινδύνου για τις αποστολές και Γίνονται τακτικές αξιολογήσεις των διαφόρων τομέων. Με υποδιέρεση κάποιες φορές ε, στις περιφέρειες κάποιου τόπου, γιατί δεν είναι έτσι ο κίνδυνος στην Κανταχάρ και σε άλλες ε, περιοχές του Αφγανιστάν. Στο Κωσυφοπέδιο δεν είναι τα πράγματα στο βορρά και στο νότο. Γίνονται λοιπόν τέτοιες αξιολογήσεις και η πολιτική ασφάλειας πλαισιώνεται στη βάση αυτή. Υπάρχουν πρότυπα ασφάλειας αποστολής τα οποία προκύπτουν από την αξιολόγηση αυτή και τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζονται. Έχουμε ξεκινήσει την εκπαίδευση των αξιωματούχων ε, σε αποστολές και πά, και ένας ε, παράγων εκπαίδευσης είναι ένα κράτος μέλος και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρεται ως ρήτρα στη σύμβαση της ε, εταιρείας. Πρόκειται για τμήμα των υποχρεώσεων του υψηλού αξιωματούχου. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, λειτουργούμε. Ίσως ο Πάτρικ θα μπορούσε να σου δώσει πιο πολλές λεπτομέρειες. Όχι. Να πω δύο λόγια μόνο για τη χρήση των πόρων των κρατών μελών. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις, σε πολλές χώρες, τα κράτη-μέλη έχουν ε, και αυτά πρόσβαση και καταφεύγουν και αυτά σε ιδιωτικέ εταιρείε ασφάλειας και αυτό καταδεικνύει πού βρίσκεται το κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό στα κράτη-μέλη. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιοι όροι για μεγαλύτερη προθυμία. Αν παρουσιαστούν αυτοί οι όροι, δεν θα τους αρνούμαστε εξ Αλλά η εμπειρία μας ως τώρα είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις οι συμβάσεις και οι ιδιωτικές εταιρείες αποτελούσαν τη μοναδική εφικτή λύση, τη μοναδική διαθέσιμη λύση μάλλον. Ρωτήσατε για τις εμπειρίες μας από συγκεκριμένε εταιρείε και καθώς υπάρχει ένας μαύρος κατάλογος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται ένα σύστημα μιας λίστας εταιριών Μια τέτοια μαύρη λίστα. Δύο στοιχεία να αναφέρω από τις πρόσφατες εμπειρίες μας. Καταρχάς αυτός ο καθολικός διαγωνισμός και διάφοροι διαγωνισμοί που έχουμε διοργανώσει στο τελευταίο, στο τελευταίο χρόνια έχουμε απομακρυνθεί από τη λογική του να διοργανώνουμε διαγωνισμούς για περιορισμένο αριθμό γνωστών ε, εταιριών. Είναι πραγματικά ανοιχτοί πλέον οι διαγωνισμοί και αυτό νομίζω ότι μας δίνει μια επιπλέον ασφάλεια ότι πραγματικά ε, δίνουμε τη σύμβαση στον καλύτερο της αγοράς. Και δεύτερο στοιχείο είναι η νέα ε, δομή της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης που είναι πάρα πολύ καινούργια. Έχουμε δημιουργήσει μια ειδική υπηρεσία, ένα ειδικό τμήμα για συμβάσεις και για διαγωνισμούς για να αντικαταστήσει την παλιά υπηρεσία προκειμένου να έχουμε επαγγελματική υποστήριξη σε ό,τι αφορά την διοργάνωση τέτοιων ε, διαγωνισμών. Και νομίζω ότι αυτό θα ενισχύσει και την ορθότητα τη στεγανότητα των πράξεών μας. Και τελευταία ερώτηση, φυσικά έχουμε μια αξιολόγηση κινδύνου τακτικά ενημερωνόμενη για όλες τις ε, χώρες και φυσικά ανταποκρίνεται στις εκάστοτε ανάγκες μας. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρος, δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Well, um, I'm sorry not to be... Και λυπάμαι που δεν είμαι πιο ακριβής. Μας εμπνέει ο κώδικας διαντολογίας και θεωρούμε ότι οι αρχές που εμπεριέχει είναι λογικές. Και γι' αυτό στις συμβάσεις μας είμαστε σε θέση να ε, συμπεριλάβουμε πολλές από τις αρχές αυτές. Ακόμα και αν από θεσμικής πλευράς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει προσυπογράψει ακόμα. If you want to... Αν θα θέλετε να προσθέσετε κάτι ακόμα, λέει ο Πρόεδρος. Well, thanks very much for... Ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε εδώ. Σας ευχαριστούμε για τις εισηγήσεις σας και ελπίζουμε σύντομα να σας ξαναέχουμε κοντά μας. Ε, πέρα στις συνεδρίασεις.